Συνάδελφοι, είναι 3 παρά 20, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε και να σας πω εδώ ότι δεν είμαι σίγουρη ότι είναι αποτελεσματικό το να αρχίζει κανείς στις 2.30 γιατί πολλοί θέλουν να φάνε και κάθε φορά που ξεκινούσαμε 2.30 αργούσαμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε λοιπόν εάν είναι χρήσιμο έτσι κι αλλιώ θα μου πείτε από την άλλη, όταν αρχίζει τρει, πολλοί έρχονται τρει και τέταρτο. Αλλά τέλο πάντων, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε. Αρχίζουμε με το σημείο 12, γύρω mapping. Γύρω mapping, λοιπόν, στα ίχνη της αναπαραγωγικής υγείας. And it's called Euromap. so now you, now you know it's item 12. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά τώρα ξέρετε πως βρισκόμαστε στο σημείο 12. Μάλλον ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο ελπίζω να ε, φτιάξουν σύντομα. Ευτυχώς. Νομίζω πως τώρα είναι όλα εντάξει. Το σημείο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η mapping είναι μια ετήσια δημοσίευση που ε, παρακολουθεί τις συνεισφορές ε, των ε, δωρητών για τα θέματα αυτά, την μητρική, βρεφική, αναπραγωγική υγεία, τον οικογενειακό προγραμματισμό. Έχουν συζητηθεί τα θέματα αυτά και στο παρελθόν, αύξηση του πληθυσμού σε πολλές χώρες, το Euro Mapping λοιπόν είναι ένα εργαλείο που χρησιμεύει στην ε, λογοδοσία και στην παρακολούθηση των δεσμεύσεων των δωρητών. Όμως έχουμε εδώ τους ε, προσκεκλημένους μας οι οποίοι είναι η Σεσίλ Βερνά από το DSW και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, EPF, από τον Neil Data. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην Σεσίλ Βερνάν για 7 λεπτά. Νομίζω πως θα μας δείξετε και ένα βίντεο μετά την παρουσίασή σας. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση. Θα είναι κοινή η παρουσίασή μας γιατί περιέχει πολλά δεδομένα και θα προσπαθήσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις αναλλαγές για να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον Ιλ για να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το έργο μας στην Επιτροπή σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπενθυμίσω γιατί είναι σημαντικό να βλέπουμε τη χρηματοδότηση ε, για την ε, υγεία των ε, βρεφών και είναι πολύ αποτελεσματική. Κάθε ευρώ που δαπανάται για οικογενειακό προγραμματισμό μπορεί να εξοικονομήσει έως και 24 ευρώ στον τομεί τη υγεία και της εκπαίδευση μεταξύ άλλων. Αυτό είναι και ο λόγος που είναι πολύ έξυπνη τακτική η επένδυση στην, ε, στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, μητρικής, βρεφικής κτλ. Να σας υπενθυμίσω ότι η χρηματοδότηση στους τομείς αυτούς σώζει ζωές γυναικών, νεογνών, βελτιώνει την υγεία, προλαμβάνει μολύνσεις με τον ε, ιό HIV, προλαμβάνει ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες μέσω του ε, οικογενειακού προγραμματισμού και βοηθά στην πρόληψη της έμφυλης βίας και της βίας κατά των γυναικών. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν ε, και όχι μόνο είναι πολύ σημαντικό να γίνονται επενδύσεις στην ε, υγεία της μητέρας και του παιδιού και την αναπαραγωγική υγεία. Τι είναι το Mapping? Είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης. Ίσως γνωρίζετε ανάλογα εργαλεία από μη κυβερνητικέ οργανώσεις το γύρο mapping λοιπόν διαφέρει γιατί λειτουργεί συμπληρωματικά. Λειτουργεί συμπληρωματικά και είναι το πρώτο που καταγράφει όχι μόνο τις δεσμεύσεις αλλά και τις εκταμιεύσεις. Παρακολουθεί τον κάθε δωρητή και την πορεία της δωρεάς, καθώς και το πόσο γενναιόδορη είναι. Ε, μεγάλες χώρες, για παράδειγμα, μπορεί να ε, κάνουν δωρεές μεγαλύτερες ε, απόλυτα νούμερα, όμως ποσοστιαία είναι ε, μικρότερες από άλλων χωρών. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ε, σε αυτό. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα, γίνεται παρακολούθηση και αυτών. Και από το 2016 η παρακολούθηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι έχει χρησιμοποιηθεί στην πολιτική, κυρίως ε, μετά την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να περιορίσει τις επενδύσεις στην αναπαραγωγική υγεία. Ε, αυτό που λέμε Global Gag Rule. Ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα, πολύ σύντομα, θα αναφερθώ στην ε, μέθοδο που ακολουθεί η Euromapping πριν δώσω το λόγο στη Σεσίλ. Ας δούμε τα δεδομένα από 30 δωρητές μέλη του ΩΣΑ. Βλέπουμε τις αιτήσιε δεσμεύσεις για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, αναπαραγωγική, μητρική, βρεφική, παιδική υγεία και ε, FP. Βλέπουμε τις αιτήσει δεσμεύσεις, αιτήσει εκταμιεύσεις και το ίδιο σε τετραετή βάση. Βασιζόμαστε στην μεθοδολογία Μουσκόκα. Μουσκόκα είναι μια πόλη στον Καναδά που το 2010 ήταν ο τόπος όπου έγιναν διεθνείς δεσμεύσεις για την βελτίωση της μητρικής και βρεφικής υγείας. Και στην σύνοδο των G20 έγιναν και επίσημες δεσμεύσεις για την ε, έβρεση κοινή μεθοδολογίας. Αυτή τη μεθοδολογία λοιπόν την πήραμε και την εφαρμόσαμε σε δεδομένα από τις χώρες δωρητές, τα οποία και αναλύουμε στην έκθεσή μας. Η Euromapping λοιπόν είναι μία άσκηση θεωρητική αν θέλετε που χρησιμοποιεί την μεθοδολογία Μουσκόκα έτσι ώστε να εντοπίσουμε την, τις ε, δωρεές για αναπτυξιακή βοήθεια στις ε, διάφορες χώρες. Και αυτό μας επιτρέπει να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη, σε αντίθεση με τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη Σεσίλ για να συνεχίσει. Προτού λοιπόν μπω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας δώσω μια συνολικότερη εικόνα της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Το 2006 λοιπόν βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν ε, ο δωρητής με τις ε, μεγαλύτερες ε, δωρεές. Η Γερμανία επίσης έχει αυξήσει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια κατά πολύ το 2016. Αν δούμε τώρα τα γραφήματα θα δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ως ε, μπλοκ, όλα τα κράτη μαζί, ε, είναι ο μεγαλύτερος δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας. Όμως, όταν πάμε στις επενδύσεις για μητρική και βρεφική υγεία, αλλάζουν τα δεδομένα. Βλέπουμε ότι εδώ οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο μεγαλύτερος δωρητής με 50%. Ε, και στο επόμενο γράφημα, πάλι αλλάζοντα ε, τον τύπο τη βοήθεια, βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ προηγούνται και πάλι με 60% ε, παρά τις, ε, τους περιορισμούς. Βέβαια, αυτό μπορεί να επιδεινωθεί. Υπάρχουν πολλές ομάδες και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες εξαρτώνται από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Και αν μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπουμε τι γίνεται με τις ε, επιμέρους επενδύσεις στη μητρική και βρεφική και παιδική υγεία. Βλέπουμε ποιες είναι οι δεσμεύσεις των χωρών για αυτό. Βλέπουμε ότι υπόσχονται, ας πούμε, δεσμεύονται να δαπανίσουν τόσα εκατομμύρια ευρώ για ε, αναπαραγωγική μητρική, βρεφική και παιδική υγεία. Και βλέπουμε εδώ ότι η Νορβηγία είναι η πρώτη χώρα που ανέλαβε πολιτικές δεσμεύσεις για ε, να διαθέσει κονδύλια για αυτόν τον σκοπό. Η Νορβηγία είναι μεν πλούσια χώρα, είναι όμως μικρή. Αναλογιστείτε λοιπόν ε, αυτό τι σημαίνει σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Μετά βλέπουμε με κίτρινο και κόκκινο τις υπόλοιπες ε, χώρες την κατάταξη των υπόλοιπων χωρών και βλέπουμε ότι οι χώρες οι οποίες έχουν ε, τις περισσότερες δυνατότητες να προσφέρουν αναψυξιακή βοήθεια είναι εκείνες που βρίσκονται πιο χαμηλά στην ε, λίστα. Τώρα, εκταμιεύσεις. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Καναδάς είναι στις ε, δύο πρώτες θέσεις. Ο Καναδάς είναι μια νέα εμφάνιση στον ε, κατάλογο αυτό. Και μετά, τρίτη χώρα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν δείτε τον κατάλογο, βλέπουμε ότι οι μεσαίες σε μέγεθος χώρες είναι εκείνες που ε, δίνουν την περισσότερη οικονομική βοήθεια. Σεσίλ, αν δούμε τώρα τις δωρές για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Βλέπουμε την ίδια τάση. Και πάλι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο μεγαλύτερος δωρητής, όμως αν μετρήσουμε την γενεοδορία της κάθε χώρας, βλέπουμε ε, να μπαίνουν στο παιχνίδι και άλλες χώρες ε, που δεν είναι ε, ισχυρές οικονομίες. Οι κάτω χώρες, για παράδειγμα, οι δεσμεύσει τους για, στον οικογενειακό προγραμματισμό είναι πολύ υψηλές. Λουξεμβούργο. Έχουν διπλασιάσει τα ποσά που διαθέτουν. Βλέπουμε λοιπόν πως αλλάζουν οι τάσεις, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις με χώρες που παραδοσιακά ε, ανήκουν ε, στην ε, κορυφή της λίστας των δωρητών, Γαλλία, Γερμανία κτλ. Εκταμιεύσεις. Εδώ βλέπουμε ότι το Λουξεμβούργο είναι στην πρώτη θέση. Πάνω από το 2,7% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας διατίθεται για ε, τον οικογενειακό προγραμματισμό και εκταμιεύεται. Δυστυχώς βλέπουμε ότι η Γερμανία, η Γαλλία και οι υπόλοιπες ισχυρές οικονομίες της Ευρωπαϊκής βρίσκονται χαμηλά. Και αυτό ίσως θα μπορούσαμε να το θέσουμε ως θέμα στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, σύνολο, βλέπουμε ότι έχει με αναλάβει δεσμεύσει για παροχή βοήθειας ε, σε όλους αυτούς τους τομείς. Υπάρχουν επίσημες δεσμεύσει στο European Consensus, στο σχέδιο δράσης ε, για τα δύο φύλλα, η πρωτοβουλία Spotlight και πράγματι βλέπουμε μια αύξηση στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά. Αρκετά μεγάλο ποσοστό τα βλέπετε κατηγοριοποιημένα αναχρώμα και βλέπουμε ότι οι επενδύσεις στην ε, αναπαραγωγική, μητρική, βρεφική και παιδική υγεία έχουν μεν αυξηθεί, όμως υπάρχει και μία στασιμότητα στον οικογενειακό προγραμματισμό. Και νομίζω πως εδώ πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα για να φτάσουμε τις πρώτες χώρες όπως το Λουξεμβούργο. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που συνεισφέρουν στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας και είναι πολύ δύσκολο να τα καταγράψουμε όλα. Αυτό κάνει και την παροχή βοήθειας ε, πιο δύσκολη. Τέλος, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι δωρητές της Ευρώπης καλύπτουν τα κενά χρηματοδότησης για οικογενειακό προγραμματισμό και αναπαραγωγική υγεία, όμως ε, βρίσκονται πίσω από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Διότι παρότι έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις δαπάνες των Ηνωμένων Πολιτείων, δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως και έπειτα υπάρχουν ελλείψεις ε, σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων. Τα δεδομένα που έχουμε παρουσιάσει είναι ήδη παροχημένα. Δεν είναι επίκαιρα, πρέπει να επικαιροποιηθούν. Μία άλλη τάση που παρατηρούμε είναι πως έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος από τις μικρές και μεσαίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις για αναπαραγωγική υγεία και οικογενειακό προγραμματισμό. Και κάποιες χώρες μάλιστα μας εξέπληξαν δεν είναι οι σκανδιναβικές χώρες που γνωρίζουμε ότι είναι πολύ προοδευτικές, όμως χώρες όπως το Λουξεμβούργο. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και η Σεσίλ, είναι μεν μεγάλος δωρητής, δεν ανταποκρίνεται πλήρως όμως στις προσδοκίες μας. Σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες ε, για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή και να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Και θεωρώ ότι με βάση τα ευρήματα αυτά ε, μπορούμε να κάνουμε πολλές ε, προτάσεις βελτίωσης. Και τώρα η Σεσίλ θα σας παρουσιάσει ένα βίντεο. Πριν δείτε το βίντεο όμως, ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι κάνει η δική σας χώρα, μπορείτε να ανατρέξετε στην έρευνά μας. Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν το βίντεο. Approximately 42 million people. So now we have the same phenomenon of tape plague. There is limited funding to the whole Uganda has a population approximately 42 million people. So now we have the same phenomenon of tape plague. There is limited funding to the whole Uganda has a population. Can we start the video again, mate? Μπορούμε να ξεκινήσουμε το βίντεο από την αρχή, παρακαλώ, και να δούμε ποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει για να το λύσουμε. Ας ξεκινήσουμε το βίντεο από την αρχή. Ευχαριστώ. Thanks, thanks, Carol. Uganda has a population approximately 42 million thanks, people thanks, with a growth rate of 3.2%. And there is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 Sorry to, I just wanted to we work with in, Λοιπόν, αυτά. Αυτό το βίντεο δείχνει τις προσπάθειες που κάνουμε ε, για την παροχή βοήθειας στους νέους ανθρώπους. Τους καλέσαμε και θα έρθουν σε μερικές εβδομάδες για να σας παρουσιάσουν την κατάσταση όπως ε, την αντιμετωπίζουν εκείνοι, την δυσκολία στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, μεταξύ άλλων. Κάνετε καλές προσπάθειες. Ναι, στις 27 Σεπτεμβρίου γίνεται μια εκδήλωση για το πώς μπορούμε να ε, βοηθήσουμε τους νέους να συμμετέχουν. Πώς μπορούν οι νέοι να κάνουν τη διαφορά, πώς μπορούν να βοηθήσουν στις ευρωεκλογές, διότι οι νέοι είναι εκείνοι που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα να σπάσουν τους ε, φραγμούς και τα εμπόδια και να βοηθήσουν. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν διάφορες ε, κοινοβουλευτικές ομάδες. Έχω μία ερώτηση για τα στατιστικά στοιχεία που έχετε. Διότι μιλήσατε για αυτό το παγκόσμιο φήμοτρο, το Global Gag. Το Νοέμβριο του 2016 εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ. Άρα λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία που έχετε από το 2016 αφορούν την ε, προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει σημειωθεί κάποια αλλαγή αν κοιτούσαμε τα στατιστικά στοιχεία τώρα που, μπορούν, που μπορεί να δείξει τις περικοπές που έχουν γίνει. Μια που μιλάμε για ε, τον Τραμπ και την κυβέρνησή του, αλλά να αναγνωρίσουμε τα στατιστικά αυτά στοιχεία είναι για, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πράγματι. Και τα στοιχεία αυτά αφορούν ε, την ε, συλλογή δεδομένων μέχρι το 2016. Και τα δεδομένα που συλλέγονται το 2017 θα αφορούν το 2016, οπότε πάμε ένα χρόνο πίσω. Τώρα, για να δούμε τον αντίκτυπο της ε, κυβέρνησης Τραμπ, ε, θα πρέπει να περιμένουμε, αλλά γνωρίζουμε ήδη ότι, υπάρχουν 30 ότι έχουν γίνει περικοπές 30 εκατομμυρίων δολαρίων στην αναπαραγωγική υγεία και επίσης ε, μείωση χρηματοδότησης, κατάργηση χρηματοδότησης για πάρα πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά, διότι δεν έχουν συλλεχθεί ακόμα. Όμως, οι νέοι περιορισμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, αν δούμε την κυβέρνηση Μπούς του νεότερου, είχαν γίνει περικοπές μόνο στον ε, οικογενειακό προγραμματισμό. Υπάρχουν διάφοροι φάκελοι, ο ένας από αυτούς είναι ο οικογενειακός προγραμματισμός. Οι διάφοροι περιορισμοί λοιπόν περιλαμβάνουν και άλλους φακέλους. Όλο το US, ε, όλη την ε, βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν αφορά μόνο τον οικογενειακό προγραμματισμό. Ο φάκελος στον οικογενειακό προγραμματισμό είχε περίπου τους 600 εκατομμυρίων δολαρίων, όμως ε, ο γενικότερος προϋπολογισμός έχει ύψος 8 δισεκατομμυρίων. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, πώς ε, διατέθηκαν τα κονδύλια, όμως το μέλλον ε, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, όπως και δεν γνωρίζουν ούτε, ούτε και στην κυβέρνηση Τραμπ, ούτε στην Ουάσιγκτον γνωρίζουν τι ακριβώς θα συμβεί. Και τι έχει χάσει η κάθε οργάνωση. Οι περικοπές έχουν γίνει σταδιακά. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε υπολογισμούς πριν έχουμε στοιχεία. Προσπαθούμε λοιπόν ακόμα να συλλέξουμε τα σχετικά δεδομένα. Η Χέιντι Χάουταλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά αυτά που μας ε, δείξατε. Πολύ σημαντικό το έργο της Euromapping. Και ε, από ευρωπαϊκής πλευράς έχουμε κάποια καλά νέα. Η Ιρλανδία, ας πούμε, που έχει αλλάξει προς το καλύτερο την ε, πολιτική της σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού. Αλλά έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αίθουσα, οπότε θα ήταν χρήσιμο πιστεύω να ακούσουμε και τι έχουν να πούν για τις δεσμεύσεις και τις εκταμιεύσεις. Αλλά, Νίλ, μας είπες ότι το τομέας αυτός έχει υπάρξει αντικείμενο πολιτικής σκοπιμότητας. και παρατηρούμε ότι κάποιες χώρες ε, διστάζουν περισσότερο από άλλες σε θέματα βρεφικής υγείας, μητρικής υγείας. Εσείς αυτό το θεωρείτε συνέπεια ε, της ε, διεύρυνσης του παγκόσμιου κανόνα, του Global Gag Rule. και υπάρχει κάποια αντιστοιχία ανάμεσα στις χώρες που χρειάζονται ε, νέα μέτρα και στις χώρες που υποστηρίζουν αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νόιζερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω στα γερμανικά για να βοηθήσω και τους ε, Γερμανούς διερμηνείς. Μάλιστα, ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τα δεδομένα που μας δώσατε. Βλέπουμε όντως μείωση ε, της χρηματοδότησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Μας το είπατε κι εσείς. Εσείς μπορείτε να κάνετε κάποιες εκτιμήσεις για το πόσο μειώθηκε η βοήθεια και κάποιες ε, προβλέψεις για το πώς ε, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντισταθμίσει τις περικοπές αυτές, αν μπορεί. Επίσης, ε, να σας πω ότι οι πληροφορίε που μας δίνετε είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την συζήτηση σε εθνικό επίπεδο, διότι εκεί ακριβώς ε, είναι το ψητό. Εκεί θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας για να δούμε τι μπορεί να κάνει κάθε χώρα στον τομέα ε, της αναπτυξιακής συνεργασίας. Και θα είναι πολύ χρήσιμο γιατί έτσι θα μπορέσουμε να πούμε, ας πούμε στη χώρα μας να κοιτάξτε τι κάνει το Λουξεμβούργο. Δεν μπορούμε να είμαστε πίσω από αυτούς. Επίσης, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση σχετικά με τις αντιδράσεις στις ε, χώρες που λαμβάνουν την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Διότι στην Ουγκάντα, ας πούμε, η άτυπη αντίδραση για τις περικοπές στον οικογενειακό προγραμματισμό από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έγιναν φυσικά δεκτές με μεγάλο ενθουσιασμό. Αλλά υπάρχουν διαφορέ. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που αυξάνει τη χρηματοδότηση, κάποια άλλη χώρα τη μειώνει τη χρηματοδότηση. Εσεί μπορείτε λοιπόν να μα ε, πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Τέλο. Μα είπατε για υπηρεσίε φιλικέ προ το χρήστη. Θα μπορούσατε να μας ε, πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό, έτσι ώστε να γνωρίζουμε κι εμείς ε, κάποια πράγματα προτού έρθουν στις 27 Σεπτεμβρίου οι οργανώσεις νέων. Ε, κυρία Σαπρόσκα έχει το λόγο. Ah, thank you. Thank you, Linda. Ευχαριστώ, Λίντα. Ευχαριστούμε πολύ τους ε, δύο μιλητές για την παρουσίαση. Θα ήθελα όμως να θέσω το εξής ερώτημα στα μέλη του πάνελ και στους εμπειρογνώμονες. Πολύ συχνά μιλούμε για το γεγονός ότι έχουν υπάρξει σημαντικές οικονομικές περικοπές και εκπτώσεις από πλευράς των εταίρων μας στις Ηνωμένες οι Ηνωμένε Πολιτείε όμω είναι μεγάλο δωρητή, παρόλο που έχουν περικόψει τη βοήθεια που δίνουν. Παραμένουν μεγάλοι δωρητέ. Και τα οικονομικά μέσα στα οποία αναφερόμαστε ισχύουν όχι μόνο στην αναπαραγωγική υγεία, αλλά και στην υγεία των νέων μητέρων, στην υγεία των νεογνών. Ε, μιλούμε για κονδύλια που προορίζονται στην φροντίδα των εγκυμονούσων γυναικών, των εγκύων γυναικών και στη βοήθεια αυτών με τον τοκητό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αρνήθηκαν να δώσουν χρηματοδότηση των αυλώσεων. Αρνήθηκαν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες δράσεις, εξ όσων γνωρίζω εκτός βέβαια των ε, καταστάσεων ε, στις οποίες ε, απειλείται η υγεία της εγγύου ή εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που η εγκυμοσύνη είναι προϊόν αιμομιξίας. Κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, η οργάνωση Μεριστούψη, η Αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Parenthood, αναφέρουν ότι παρέχονται και άλλες υπηρεσίες υγείας. Δεν περιορίζουν την υπηρεσία τους στο να προσφέρουν αμβλώσεις μόνο. Ανησυχούν όμως ότι θα μειωθεί η χρηματοδότησή τους στο μέλλον. Και αυτές οι οργανώσεις θέλουν να τη χάνουν χρηματοδότησης από την ε, κυβέρνηση των ΗΠΑ. Επομένως, γιατί επιμένουν να παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο με αμβλώσεις που να έχουν να κάνουν μόνο με τέτοιου είδου δράσεις και γιατί δεν διευρύνουν ε, το, την πληθώρα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα, έχουν, ε, δεν θα υφίστανται αυτό το κίνδυνο του αποκλεισμού τους από τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Πολλά είναι τα ερωτήματα, παρακαλώ. Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ τα αξιότιμα μέλη για τις ερωτήσεις τους. Πρώτον για την ε, πολιτικοποίηση και αυτά που είπε η κυρία Χάουταλα. Είναι ένα θέμα που έχει αποκτήσει μεγάλες πολιτικές διαστάσεις. Έχει γίνει πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Κάποιες οργανώσεις κινδυνεύουν να χάσουν την ε, χρηματοδότησή τους και γι' αυτό κάποιοι είναι διστακτικοί. Δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη ΣΥΠΑ για συγκεκριμένα ζητήματα. Υπάρχει δηλαδή μια ντροπαλότητα, ένας δισταγμός, μια επιφυλακτικότητα γιατί το θέμα έχει αναχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα στις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν θέλουν να υπονομευτεί η χρηματοδότησή τους λόγω αυτού. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις γειτονικέ χώρες και τη θέση τους για τον οικογενειακό προγραμματισμό μεταξύ άλλων είναι το ότι οι δωρητές στηρίζουν με πολλά και διαφορετικά επίπεδα από τη μία χώρα στην άλλη ή από τη μία χρονιά στην άλλη. Στις Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν στροφή 180 μοιρών αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη. Δεν μπορεί κανείς να, να πει ότι δεν φταίμε σε τίποτα, γιατί οι παραδοσιακοί δωρητέ έχουν τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο δίνουν τη χρηματοδότηση και αυτό έχει επηρεάσει τις χώρες υποδοχή που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση. Σε αυτέ τι χώρε αυξάνεται η πολιτική στήριξη σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα του οικογενειακού προγραμματισμού. Είχαμε τις πρώτες θετικές ε, ε, υποδοχές του προγράμματος τις αρχές του 2010, περίπου το 2012 δηλαδή, και στη συνέχεια έχουμε εξαπλώσει την δράση μας και σε νέα πεδία. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, Ποιε είναι οι επιπλοκέ των περιορισμών των κονδυλίων. Τι θα γίνει δηλαδή αν αποκλειστικά και μόνο ε, παίρνουμε κονδύλια από το EDPPF. Νομίζω ότι έχετε παρανοήσει κάτι. Κάτι που πρέπει όλοι να γνωρίσουμε για τη χρηματοδότηση των ήπα είναι το εξής. Οι ήπα είχαν νόμιμη απαγόρευση της χρηματοδότησης των αμβλώσεων σε τρίτες χώρες από το 1973. Δηλαδή από το 1973 η χώρα αυτή έχει απαγορεύσει να χρησιμοποιείται χρηματοδότηση δική της για σκοπούς αμβλώσεων σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Υπάρχει ειδικό νόμος του Κογκρέσου από το 1973. Όμως αυτό το συγκεκριμένο που έκαναν τώρα ήταν να μην χρηματοδοτήσουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες ε, λαμβάνουν χρηματοδότηση για κάποια ζητήματα και κάνουν και αμβλώσει παράλληλα για τις οποίες δεν χρησιμοποιούν την αμερικανική χρηματοδότηση αλλά χρηματοδότηση από άλλες χώρες. Επομένως, εάν μια γυναίκα επισκεφτεί μια κλινική και θέλει άμβλωση και δεν την παρέχει και αν πει η μη κυβερνητική οργάνωση, «Ε, εμεί εδώ δεν κάνουμε αμβλώσει πρέπει να πάτε στο τάδε μέρος, αυτό σχετίζεται με την άμβλωση και αν το χρηματοδοτεί αυτή την ώρα του υπαλλήλου άλλο ο δωρητής, τότε αυτή η οργάνωση πάβει πλέον να είναι επιλέξιμη να λάβει η Αμερικανική χρηματοδότηση μόνο και μόνο επειδή έδωσε οδηγίες για το πού γίνονται. Άρα, να είμαστε σαφείς. Είναι κάτι που υπάρχει για περισσότερο από 40 δεκαετίες και ε, έχει να κάνει με αμερικανικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες για το θέμα των αυλώσεων δέχονται πορού από άλλε πηγές. Χάνουν την επιλεξιμότητά τους για τι αμερικανικές πηγές χρηματοδότηση και αυτό ε, ισχύει ανεξαρτήτως από το κατά πόσο είναι νόμιμες και λειτουργούν νόμιμα. Σε πάρα πολλές χώρες η άμβλωση επιτρέπεται υπό ορισμένε περιπτώσεις, βεβαίως πολύ περιορισμένες συγκριτικά με την υπόλοιπη την Ευρώπη, αλλά στις περισσότερες χώρες της Αφρικής είναι νόμιμη ή είναι δυνατή η άμβλωση για να σωθεί η υγεία της μητέρας. Και θα χάσουν τη χρηματοδότηση αν ασχοληθούν. Ε, Περί αυτού πρόκειται. Δεν πρόκειται για τη χρηματοδότηση των αμβλώσεων. Είναι κάτι που υπάρχει και ισχύει για πάντα από 40, από 4 δεκαετίες. Να συμπληρώσω το εξής. Θέλουμε οι γυναίκες να κάνουν ενημερωμένες επιλογές, να τις ενημερώσουμε για τα δικαιώματά τους και για τις δυνατότητες τους. Και θέλουμε ακριβώς να αποφύγουν την άμβλωση να μην καταλήξουν να φτάσουν στο σημείο να χρειάζονται άμπλωση και αυτά είναι τα project που κάνουμε στη Κένια. Ε, θα πρέπει να έχουμε στοιχεία και προφορίες. Πολλές είναι οι οι επιπλοκές, αν θέλετε, και οι διακλαδώσεις αυτού του θέματος. Στην Επιτροπή μας υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και τίθεται το θέμα. Πώς αυτά θα τα εξορροπήσουμε με αυτό που γίνεται σε χώριο επίπεδο. Έχουμε δεσμεύσεις, έχουμε γραμμές του προϋπολογισμού, στην Κένια και στην Ανατολική Αφρική έχουμε γραπές του προϋπολογισμού για τον οικογενειακό προγραμματισμό, όμως στην εφαρμογή τα κενά είναι πολλά και διάφορα. Δεν υπάρχει αρκετή πρόσβαση σε βασικά αγαθά, π.χ. στην Κένια. Όλα αυτά έχουν κάνει και με την αποκέντρωση, όλα γίνονται σε τοπικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο συχνά απουσιάζουν δεξιότητε δεξιότητες και οι ικανότητες για τη διαχείριση όλων αυτών. Πολλά λοιπόν πρέπει να βελτιωθούν στο ε, τομέα της εφαρμογής. Το ίδιο ισχύει και για την νεολαία η οποία έχει αναγνωριστεί ως προτεραιότητα για τις χώρες αυτές, τις περισσότερες από αυτές τις χώρες, γιατί είναι πολύ μεγάλη δυναμική ε, μεταβολών στο πληθυσμό. Όμως, σε ό,τι έχει να κάνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες για χαθά από πλευράς νέων, δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση. Δεν είναι οι υπηρεσίες αυτές εμπιστευτικέ. Δεν μπορεί ένας νέος, για παράδειγμα, να βρει πληροφορίες για τη σεξουαλικότητα, για διάφορα θέματα, χωρίς να περάσει από την νοσοκόμα η οποία γνωρίζει προσωπικά τους γονείς αυτού του νέου ή της νέας, για παράδειγμα, και θα τα μεταφέρει. Και γι' αυτό υπάρχουν δισταγμοί και προβλήματα όλα αυτά τα πρότυπα μπορεί κανείς να τα αναπτύξει, να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματίες της υγείας γνωρίζουν αυτά τα πρότυπα και τα εφαρμόζουν, είναι μια σειρά από μικρά βήματα που γίνονται για να έχουν οι νέοι πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα. Και είδατε στο βίντεο ότι όλοι νέοι που μίλησαν θέλουν και έχουν γίνει σιγά σιγά όλοι οι ακτιβιστές υπέρμαχοι αυτού του σκοπού. Και κάνουν αλλαγές στη ζωή τους και στην υπόλοιπη κοινωνία. Θα δούμε και το θέμα της Τανζανίας, θα έχουμε σχετική εκπρόσωπο που έχουμε προσκαλέσει για το Σεπτέμβριο. Από τον κύριο Είχαμε την ερώτηση για το τι γίνεται με την αντιστάθμιση από τους Ευρωπαίους δωρητές και τι γίνεται με τις ε, πιθανές ε, απώλειες ζημίες από τη ΣΥΠΑ. Τώρα θα πρέπει να επεκταθεί ε, ο κανόνας του φήμωτρου και τώρα έχουν αφιερώσει πολλά χρηματοδότηση ώστε να αντισταθμιστεί η απόλυτη της Αμερικανικής χρηματοδότησης. Αυτό είναι τον. Φεβρουάριο με Μάρτιο του 17 Και είναι πάνω από 400 εκατομμύρια. Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Βέλγιο, Κατοχώρες, Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο συνέβαλε. Και το Λουξεμβουργείο. Το Ηνωμένο Βασίλειο με κάπως διαφορετική μέθοδο. Οπότε αντέδρασε η διεθνής κοινότητα. παρόλα αυτά νομίζω ότι τόσα πολλά προγύπτουν τώρα από πλευράς Αμερικής που είναι κατά της διεθνούς τάξεως που δεν είναι τόσο μεγάλο κίνητρο το τι κάνει η Αμερική για τους Ευρωπαίους δουλείτες που περισσότερο ενδιαφέρονται για να υπάρχει οικογενειακός προγραμματισμός με αυτόν τον τρόπο που είναι το σωστό. Πρόεδρος, να δώσουμε το λόγο ξανά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλουν να πούν κάτι. Κέβιν Μακάρτη. Από την ΔΕΒΚΟ, από την υπηρεσία που ασχολείται με την υγεία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Και ευχαριστούμε μας για την ευκαιρία να σχολιάσουμε. Βεβαίως και θέλουμε πολύ τις προσπάθειες του φορέα αυτού, του DSW. Και αποδεχόμαστε τον έλεγχο από πλευρά του. Θα πρέπει και εμεί να είμαστε των περιστάσεων. Θα πρέπει να είμαστε πρωτότυποι όσον αφορά την προσβασιμότητα γυναικών, μεγάλων και μικρών. Ε, να μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων τους με ισότητα και αυτά αποτυπώνονται στα έγγραφα πολιτικής για το πρόγραμμα δράσης, για τα δύο φύλλα κλπ. Έχουμε πάρα πολλά μέσα πολιτικής, γεωγραφικά, παγκόσμιες πρωτοβουλίες, με συνεργασία με το ΝΟΙΕ, UNFPA, οπότε και για, το, για τη μέθοδο αυτή έχουμε δώσει πάρα πολλά χρήματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο πέρσι και έχουμε αυτήν την ε, πρωτοβουλία. Περιμένουμε ακόμη περισσότερη στήριξη από το Κοινοβούλιο όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε ε, την ε, στρατηγική μας για τη μέθοδο αυτή μέσω των συνομιλίων που τώρα προχωρούν. το 2017. Επομένως ε, είχαμε πάρα πολλές ε, δαπάνες που αφορούσαν ε, αυτή την υπόθεση της υγείας και περίπου 30% αυτής της χρηματοδότησης πήγε σε αυτά τα θέματα προγραμματισμού και υγείας. Και ευχαριστούμε αυτούς που διοργάνωσαν την σημερινή συνάντηση και βεβαίως θα πρέπει να δούμε τι προτεραιότητες έχουν ε, τεθεί και να ξέρουμε από πλευρά αναπτυξιακή πολιτική τι προβλέπεται. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε και μα τα παρουσιάσατε όλα αυτά που ενδιαφέρουν την ε, Επιτροπή μας. Σα ευχαριστούμε. Okay. Yeah, we're going to move on to item 13. We're going to back... Προχωρούμε τώρα στο 13. Περιμένουμε να έρθει ο κύριος Αμιλάτ. Περάστε, καθίστε. Προχωρούμε στο 13, Αυτό το σημείο αυτό αφορά την συνεργασία με το Ιράν, δυνάμει του μέσου ανοιξιακής συνεργασίας, του DCI. Εδώ έχουμε τον κύριο Αμιλάτ όσον αφορά τα θέματα συνεργασίας, διευθύντη, συνεργασία με Ασία και άλλε περιοχέ. Και αυτά όλα μα αφορούν διότι το καλοκαίρι ε, ε, αποφάσισε να υπάρξουν ειδικά μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτή, στα πλαίσια αυτά έχουμε 18 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε στα πλαίσια αυτά 8 εκατομμύρια για τεχνική βοήθεια, 8 εκατομμύρια για το περιβάλλον, νερό, έδαφος ε, κλπ. Και, και 2 εκατομμύρια για ζητήματα υγεία για όσους είναι οροθετικοί, πάσχουν από έτσι τέλος πάντων και όλα αυτά προχώρησαν ε, ταχαίως. Ίσως θα θυμάστε ότι τον Μάρτιο πέρσι είχαμε τον στατικό διάλογο με τον Επίτροπο Νίμτσα και μας έλεγε ότι δεν είχε υπόψη του κάτι σχετικό ε, και αυτό δεν άρεσε στους συναδέλφους, δηλαδή το θέμα συνεργασίας με το Ιράν, αλλά ε, είναι γνωστό το πόσο σημαντική υπόθεση είναι ε, το να υπάρχει κάποια συμφωνία και συνεργασία με το Ιράν. Ο προχωρήσαμε προς αυτήν την κατεύθυνση της συνεργασίας με το Ιράν και στις 19 Ιουλίου η γραμματεία μας ειδοποιήθηκε ότι θεσπίστηκαν αυτά τα ειδικά μέτρα. Ταχύως. Συμφωνήθηκαν. Όμως έτσι όπως το έκαναν, δεν δείχνουν πρόβλημα συνεργασίας. Δεν σεβάστηκαν το ελεγκτικά, τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Είχαμε το πολιτικό φόρμ του επίπεδου τον Ιούλιο. Αλλά βέβαια είναι γνωστό ότι όταν το Κοινοβούλιο έχει διακοπή λειτουργίας δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες του. Επομένως θα πρέπει να μας εξηγηθεί γιατί προχώρησε σε τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιουλίου είπαν στα κρατημέλη ότι όλα αυτά θα κρυθούν και οριστικά με λήφθη απόφαση στις 19 Ιουλίου. Και το φθινόπωρο θα προχωρούσε ακόμη περισσότερη υπόθεση. Αλλά μόνο τότε θα μπορούσε να συζητηθεί η ουσία του θέματος. Γιατί έγινε αυτό, γιατί πρέπει να γίνει κατά τις διακοπές. Δεύτερον, γιατί ως μέσον επελέγει το DCI, ενωτησιακή συνεργασία. Έχουμε 8 εκατομμύρια για το εμπόριο. 8 εκατομμύρια για την ε, ρήπανση των υδάτων και 2 εκατομμύρια για την υγεία. Ξέρουμε ότι το Ιράν είναι μια χώρα με εισοδήματα μεσαία προς υψηλά δεν είχε πριν ε, κάλυψη από ορδιπισιακά μέτρα. Μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέτρα. Άρα πολλά είναι τα ερωτήματα. Γιατί διαλέξατε αυτά τα μέτρα και μετά να δώσουμε το λόγο στην Σεσίλ που είναι επικεφαλής της ομάδας ελέγχου κύριος Αμιλάτο όμως, πρώτος να λάβει το λόγο. Να μας εξηγήσει. Σεσίλ, στη συνέχεια εσύ θα λάβεις το λόγο. Για να μας εξηγήσεις τι δυσκολίες ε, είχες όσον αφορά την παρατήρηση των εκλογών στο Μαλί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε και να σας εξηγήσουμε και να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν γίνει γραπτά. Στείλαμε μια γραπτή απάντηση λοιπόν. Νομίζω πως ε, λάβατε την απάντηση από τον Επίτροπο Μίμητσα. Και μάλιστα μέρος της απάντησης επαναλαμβάνει αυτά που είχαμε πει εν είδη εξήγηση στα πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου για την ενδιάμεση αξιολόγηση της ε, βοήθειας και για τις προτάσεις που είχαν γίνει την εποχή εκείνη για διμερείς ε, συνεργασίες με το Ιράν. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια δυνατή πολιτική ε, πλατφόρμα ε, για, αυτά, για ό,τι κάνουμε με το Ιράν, για όποια συνεργασία έχουμε. Δεν ε, δρούμε αυθαίρετα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα θεσμικά της όργανα, με τα κράτη-μέλη συμμετέχουν πλήρως. Και στις 27 Μαΐου τα κράτη-μέλη ενημέρωσαν εκ νέου για την στήριξή τους. Ήταν πολύ μεγάλη απόφαση. και την έγκριση μέτρων για την υποστήριξη όχι μόνο ευρωπαϊκών φορέων αλλά και για την συνέχιση της ε, τομεακής συνεργασίας με το Ιράν και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Αυτό μόνο προκάλεσε την ε, ανάγκη για ε, εξακολουθητική δράση. Και όπως γνωρίζετε, για να έχεις αποτελέσματα υπό τέτοιες συνθήκες πρέπει να εργάζεσαι πάρα πολύ γρήγορα, με επισπεσμένες διαδικασίες. Η ταχεία λοιπόν έγκριση των μέτρων αυτών ήταν αποτέλεσμα ε, πολιτικής βούλησης στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν. Και φυσικά υπήρχε και διεθνές ε, πολιτικό κλίμα πρόσφορο, με δηλώσεις, με απόσυρση επενδύσεων από τη χώρα, Αυτό λοιπόν οδήγησε τα κρατημέλη αλλά και τα θεσμικά όργανα να ασκήσουν πίεση στην Επιτροπή για να έχει αποτελέσματα ταχύτερα. και να τηρήσει τις ε, διάφορες δεσμεύσεις που έχουν γίνει. Αυτό νομίζω πρέπει να το θεωρήσουμε ως ε, ένα μήνυμα το οποίο βέβαια είναι λυπηρό ότι εδόθη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όλα αυτά βέβαια δεν έχουν ε, δεν σημαίνουν μάλλον ότι εμείς ε, δεν λογαριάζουμε το Κοινοβούλιο και το δικαίωμά του για κοινοβουλευτικό έλεγχο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, στην οποία αναφέρεστε, για κράτη-μέλη τα οποία ενημερώνονται μία εβδομάδα πριν, να σας απαντήσω ότι τα έγγραφα στάλθηκαν ταυτόχρονα στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη. Και οι πληροφορίες αυτές υπήρχαν. Δεν ε, Δείξαμε λοιπόν προτιμησιακή συμπεριφορά σε ορισμένα κρατημέλη, σε όσους ήταν παρόντες δηλαδή. Σίγουρα λοιπόν ο έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός για εμάς. Ε, ερχόμαστε με μεγάλη χαρά εδώ για να σας ενημερώσουμε και σας ε, διαβεβαιώνω ότι θέλουμε να σας ενημερώνουμε, θέλουμε να σας κρατούμε ενήμερους. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες στις συμφωνίες ε, με το Ιράν και σίγουρα το όλο θέμα αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Έχουν εγκριθεί λοιπόν ειδικά μέτρα με επισπεσμένη διαδικασία. Εγκρίθηκαν στις 27 Αυγούστου και υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσαμε να έχουμε ε, ξεπεράσει το πρόβλημα το, της θερινής διακοπής λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Όμως, ακριβώς επειδή ο χαρακτήρας ήταν κατεπήγον και έπρεπε να σταλεί αυτό το πολιτικό μήνυμα, αναγκαστήκαμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Σας στείλαμε λοιπόν μία περιγραφή της ε, δράσης, μία πλήρη περίληψη, ε, ουσιαστική, και παραδεχόμαστε ότι έγινε ένα μικρό λάθος που αφορά την ε, συμπερίληψη του κειμένου και γι' αυτό σας ζητώ και σήμερα συγγνώμη. Και νομίζω πως η απάντηση στις ερωτήσεις σας είναι η ουσία αυτών που έχουμε απαντήσει. Να σας υπενθυμίσω ότι τα μέτρα εστιάζουν σε τομείς συνεργασίας ε, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, όχι μόνο για το Ιράν, αλλά και για εμάς και για όλη την περιοχή. το η κατάσταση περιβαλλοντική στο Ιράν είναι άθλια. Το Ιράν ε, ζει την χειρότερη ξηρασία εδώ και 50 χρόνια. Η ρήπανση στις πόλεις είναι ε, πολύ υψηλή. Υπάρχουν ε, θύελες σκόνης που καταστρέφουν ομάδες πληθυσμού, χωριά. Τώρα, χρήση ναρκωτικών. Προσοχή, εδώ μιλάμε για χρήση, για κατανάλωση, όχι για ε, κάτι άλλο. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίω. Θεωρείται ότι ότι το 90% των ναρκωτικών ουσιών περνά από το Ιράν. και η χρήση δυστυχώς πλήττει πολλούς ε, κατοίκους της χώρας. Αυτό συνδέεται και με την ε, μόλυνση από διάφορες ασθένειες, όπως για παράδειγμα από τον HIV. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το οικονομικό για τη χώρα. Το νόμισμα του Ιράν έχει χάσει το ίμιση της αξίας του το τελευταίο εξάμεινο υπάρχουν πολλοί που έχασαν όλες τους τις οικονομίες και η χώρα είναι στο χείλος της οικονομικής καταστροφής δεδομένων και των οικονομικών κυρώσεων που θα επιβληθούν σύντομα. Όλα αυτά αναφέρονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2016. Αν δείτε το ψήφισμα, προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι όλα αυτά που προτείνουμε ε, γραπτός, όλα αυτά τα μέτρα, αφορούν τομείς οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, πολύ σημαντικοί. Είναι τομείς όπου υπάρχει ανάγκη για δράση. Εσείς οι ίδιοι το έχετε πει. Επίσης, δεν αναφερόμαστε ρητά στις ναρκωτικές ουσίες, διότι όπως γνωρίζετε στο Ιράν ε, υπάρχει ακόμα η θανατική ποινή και δεν ε, θέλαμε να ε, δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουν χαλαρώσει, έχει χαλαρώσει κάπως η νομοθεσία σχετικά με τη θανατική ποινή και αυτό πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, πέρα από αυτά τα μέτρα, να είμαστε ενεργοί σε θέματα ε, μετανάστευσης, ε, εκτοπισμένων πληθυσμών. Όπως ξέρετε, υπάρχουν 3 εκατομμύρια Αφγανοί στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τεράστια ανάγκη στήριξης των ανθρώπων αυτών. Επίσης, στηρίζουμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Ιράν. Και σε ό,τι αφορά τη χρήση των μέσων αυτών, το μέσο για την εταιρική σχέση δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τομείς της συνεργασίας, μόνο σε ορισμένους. και δεν έχει τόσο ε, μεγάλη χρηματοδότηση όσο άλλα, όπως ε, το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Εκεί πρέπει να δοθεί ίσως έμφαση διότι πολλά μέτρα έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα και αφορούν για παράδειγμα διαχείριση υδάτων, αποβλήτων, ε, μόλυνση στην Κασπία θάλασσα που διαχειρίζονται οι αρχές του Ιράν. Και είναι προς το συμφέρον όλων να βοηθήσουμε και εμείς. Επίσης, οι προϋποθέσεις που θέτει το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας για πρόσβαση στη χρηματοδότηση νομίζω πως ε, εξηγούν επαρκώς ε, τις ε, ενεργειές μας. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν απαντήθηκαν όλα μου τα ερωτήματα. Η Επιτροπή για το Μέσο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία συνεδριάσε τον Ιούλιο και είχε μάθει ότι θα έχει τα έγγραφα τις επόμενες εβδομάδες και η δική μας Επιτροπή συνεδρίασε στις 11 Ιουλίου. Δίνουμε στην Επιτροπή το λόγο στην αρχή κάθε φορά για να μας πει τι θέλει να θέσει. Εγώ ήμουν με τον Επιτρόπο Μίμητσα στη Νέα Υόρκη και είδαμε αξιωματούχους από την DJ Τεύκο και κανείς δεν μου τίποτα. Μετά που γύρωσα ε, πήραμε το σημείωμα το τσέκαρα και το, ξανα... το διπλό τσέκαρα. Αποφασίσαμε το Μάιο και τελικά στις, στις 6 Αυγούστου πρόκειται να ε, ε αυτά τα μέτρα. δεν νομίζω ότι αποφασίσατε αυτά στις 11 Ιουλίου ότι ήταν το επίγον. Τα ξέρετε από πριν και δεν τα είπατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να μας εμπλέκετε. Να δώσω το λόγο στη Σεσίλ Κέγκε που χρειάστηκε να το χειριστεί το θέμα. Σεσίλ, παρακαλώ. Είναι πρόεδρος της ομάδας κοινοβουλευτικού, κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ευχαριστώ, Λίντα. Νομίζω ότι πολλές ερωτήσεις έχουν ήδη τεθεί και θα προσπαθήσω να κάνω μια χρονολογική ε, αναδρομή στα γεγονότα και θα προσπαθήσω να θέσω κάποια ερωτήματα. Αλλά υπάρχουν κι άλλα. Και σε κάποια έχει απαντήσει ο κύριος Αμίλα. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 19 Ιουνίου η Γραμματεία δεχόταν δύο έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίληψη και παράρτημα για σχέδιο ειδικά μέτρα για το Ιράν 18 εκατομμύρια ευρώ σε τρία σκέλη. Τα τρία αυτά σκέλη μας εξηγήθηκαν από τη Λίντα και από τον κύριο Αμιλά. 8 εκατομμύρια ευρώ τεχνική βοήθεια για τις εμπορικές ανταλλαγές, στήριξη μικρομέσων επιχειρήσεων, βελτίωση της ε, αλυσίδας ε, αξιών, ε, κάποια εκατομμύρια επίσης για την καταπολέμηση της ρήπανσης του νερού και του αέρα, για την καταπολέμηση της υποβάθμισης των εδαφών και για την ενίσχυση της διαχείρισης των αποβλήτων και 2 εκατομμύρια ευρώ για ειδικέ ανάγκε για την περίθαλψη, για την υγεία, για του ασθενεί από, από τον ιό HIV, AIDS, ε, για ε, τους ναρκωμανείς και το καθεξής. Είχαμε γραπτή διαδικασία με καταληκτική προθεσμία 31 Ιουλίου. Αυτό το ειδικό μέτρο ε, το ενημερώσατε το Κοινοβούλιο στο τέλος της ε, τυρκουάς εβδομάδας του Ιουλίου και τις παραμονές των διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς τελικά ε, το θεωρούμε ότι μας ενημερώσατε σε ένα τέτοιο δύσκολο χρονικά σημείο ακριβώς γιατί θελήσατε να στερήσετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα νόμιμα δικαιώματα κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχει. Δεν ήμουνα εδώ γιατί είναι σε εβδομάδα τυρκουάς και ήμουνα σε αποστολή και δεν έπρεπε να βρίσκομαι εδώ και γι' αυτό δεν ήμουνα. Και δεν μπόρεσα να εργαστεί η αρμόδια ομάδα εργασίας κατά τη διάρκεια των διακοπών του Αυγούστου. Και έπρεπε να εγκριθούν όλα αυτά με τη γραπτή και σιωπηρή διαδικασία πριν σταλούν στην Πρόεδρο και στον Επίτροπο Μίμητσα στις 30 Ιουλίου. Δεν έγινε έτσι ο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτά κάνατε εσεί, αλλά δεν μπορεί να έτσι να γίνει. Και έχουμε ειδικά μέτρα αντίθετα και εκφράζουμε τη θέση μας και θέλουμε η θέση μας να διαβαστεί στα κράτη-μέλη. Επομένως, η Επιτροπή μας, η ΝΤΕΒΕ, δεν αγνοεί το πολιτικό πλαίσιο, το οικονομικό και διαπληματικό πλαίσιο των λανθάνων, ε, των περιραίων. Δεν αγνοεί τη Σύνοδο της Σόφιας της 17ης Μαΐου. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και αποφάσισαν να προσχωρήσουν σε αυτή όπως το Ιράν και να τηρήσουν πλήρως τη δεσμεύσεις από τη στιγμή που το δύο θα κάνει και αυτή η χώρα. Αναγνωρίζουμε ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε τις αντιδράσεις των κρατών μελών στις αρχές Αυγούστου ή στα μέσα Αυγούστου και το γεγονό ότι επανενεργοποιούνται οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν είναι θλιβερό. Ε, η Επιτροπή μας ε, λυπάται γιατί δεν μπόρεσε να ασκήσει τα δικαιώματά της για το κοινοβουλευτικό δημοκρατικό έλεγχο για τα ειδικά μέτρα που λήφθηκαν. Επομένως, με αυτή τη χρονολογική αναδρομή στα γεγονότα καταλαβαίνει κανείς ότι μια πιο στενή συνεργασία θα ήταν προτιμότερη. Αυτά τα ειδικά μέτρα όμως που επανανεργοποιήθηκαν και ξανατέθηκαν σε ισχύ θα έπρεπε να τύχουν ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεδομένου του γεγονότο ότι ήδη έχει αποφαθεί για το θέμα αυτό το Κοινοβούλιο στο παρελθόν, αλλά και ε, ε, με την ευκαιρία του στρατηγικού διαλόγου για την ε, εξέταση και την ενδιάμεση αναθεώρηση των σχετικών εγγράφων, τον Μάρτιο ε, το Κοινοβούλιο είχε απευθύνει επιστολή στον Επίτροπο Μίμητσα και είχε εκφράσει επιφελάξεις για τον διμερή ε, καταμερισμό ε, για το γεγονός ότι έχουν τεθεί κατά μέρος τα 50 εκατομμύρια ευρώ για το Ιράν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μας εξού και υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης του ειδικού αυτού μέτρου ενώ απουσιάζουν οποιαδήποτε έγγραφα πολιτικής και προσανατολισμού για το Ιράν. Ο Επίτροπος, ο Επίτροπος Μίμητσα μα ενημέρωσε ότι τη θέση μας την έχει διαβεβάσει στα κράτη-μέλη πριν από τις 31 Ιουλίου και επρόκειτο να ενημερώσει τα κράτη-μέλη που ήταν υπέρ και ο σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοθέτηση ειδικού μέτρου για το Ιράν και όταν θα γίνει η ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμματικών εγγράφων μέχρι τις 20 Ιουλίου. Αυτό ήταν η συνολική ευκαιρία να δοθούν 50 εκατομμύρια ευρώ για το Ιράν. Έχουμε ήδη εκφράσει επιφυλάξεις το Μάρτιο και οι επιφυλάξεις μας έχουν καθησυχαστεί για την περίοδο 2018-2020. Το ειδικό μέτρο για το Ιράν έτυχε έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν σημεία που ήθελα να υπογραμμίσω στην παρέμβασή μου και τα οποία ήδη έθιξε ο κύριος Αμιλά, μεταξύ άλλων. Άρα δεν χρειάζεται να επεκταθώ περαιτέρω, μπορώ να απαντήσω και σε ερωτήσεις για όλη αυτή τη διαδρομή. Πρόθεση μου όμως είναι να τονίσω ακριβώς αυτό. ότι δεν επιτράπει στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές να ασκήσουν το κοινοβουλευτικό δικαίωμα ελέγχου και έκφρασης που διαθέτουν. Όμως, το γεγονός δεν έγινε αυτό δεν σημαίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η κοινοβουλευτική διαδικασία. Έγινε αυτό γιατί έλειπαν όλοι οι διακοπές. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέσω της γραπτής διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη Σεσίλ γιατί μας έδωσε τις λεπτομέρειες και το χρονολογικό υπόβαθρο. Τρεις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο Σάρλ Γκέρεντς, η κυρία Χαουτάλα και ο κύριος Σαφχάουσερ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Σάρλ, παρακαλώ. Σειρά σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια διότι με διάβγεια και σαφήνεια παρουσίασε το ιστορικό χονοδριά, χονοδιάγραμμα αυτών των δράσεων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης άκουσα να γίνεται λόγος για το Ιράν, της ενδιάμεσης αναθεώρησης του προγράμματος που έχουμε για την ευρύτερη περιοχή. Και τότε είχα απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την είχα ρωτήσει συμφωνούν αυτά με την αρχή της διαφοροποίησης. Και εξ όσων κατάλαβα και αν δεν απατώμε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, και ερμηνεύω βεβαίω τα λόγια του ενδεχομένω λάθος, ότι ε, είπαν λοιπόν ότι η αρχή της διαφοροποίησης είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαταλείπει σιγά σιγά. Προσωπικώς δεν έχω πρόβλημα με αυτό, δεν με ενοχλεί να το πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Γιατί αν εντάξουμε την ε, αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, προοπτική της μείωσης των ανισοτήτων σε όλες τις χώρες, που είναι θεμητός ε, σκοπός και μάλιστα στις χώρες ενδιάμεσου εισοδήματος, τότε πρέπει να θετήσουμε μια πολιτική που να αποστασιοποιηθεί από την αρχή της διαφοροποίησης. Γιατί η αρχή της διαφοροποίησης είναι που τους είχε αποκλείσει. Καλώς λοιπόν, άριστα ω προς αυτό. Δεύτερον, Επίσης καταλαβαίνω και κατανοώ το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει, επιδιώκει, αποσκοπεί να έχει θετική απήχηση σε μια χώρα η οποία δημιουργεί προβλήματα και η οποία δημιουργεί προβλήματα γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, διαρρήξει τις ε, σχέσεις συμφωνίας που έχουν με αυτή τη χώρα. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω και τα κατανοώ. Να μας ενημερώνετε όμως για τις πολιτικές επιλογές οι οποίες ε, δίνουν λαβή για να δοθεί άλλη ερμηνεία σε αρχές οι οποίες είναι δικές και και οι οποίε έχουν εγκριθεί με τη δική μα συμφωνία ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, αυτό θα πρέπει να το πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην αφήνει να εξαφανίζεται σε θολά νερά σκέλο τη Ευρωπαϊκή Πολιτική και των ευρωπαϊκών αρχών. Δεν είναι σωστή αυτή η άγουσα για του νέου μελλοντικού προσανατολισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο ερωτήματα, δύο ζητήματα τώρα πιο τεχνική φύση ε, θα ήθελα να θέσω. Να συμφωνήσουμε εδώ ότι δεν έχουμε προσέγγιση ως προς τη βοήθεια προς το προϋπολογισμό, αλλά έχουμε προσέγγιση ανα project, ανα πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι. Αυτό καταρχάς. Και δεύτερον, τι γίνεται με τις άλλες χώρες και με χώρες τύπου Ιράν. Με χώρες με τις οποίες δηλαδή θέλουμε να διατηρήσουμε κάποιες σχέσεις ε, σε ένα κάποιο επίπεδο. Δηλαδή να διατηρήσουμε το διάλογο να, να προλάβουμε να μην γίνουν παρεκκλήσεις και να μην ε, ε, εκτραχυνθούν και ξεφύγουν τα πράγματα. Να διατηρήσουμε κάποιες τυπικές σχέσεις δηλαδή δεν θα ήταν σκόπιμο και φρόνιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί επί της αρχής πώς θα αντιμετωπίζει τις χώρες αυτές, θα ενθαρρύνει τις εκλεγμένες κυβερνήσεις ή τις επέσπιπτος υφιστάμενες κυβερνήσεις ή θα τις θεωρήσει υπεύθυνε. Στα λόγια του Διευθυντή Αζή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανείχνευσα και τις δύο ε, επιλογές. Όμως στα μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα, όταν θα τα προσδιορίσουμε και θα τα αποφασίσουμε, θα πρέπει να συζητήσουμε και για τις αρχές και να έχουμε πιο ξεκάθαρη άποψη για τα κατά πόσο είναι έγκυρες οι πολιτικές μας. Αυτά λοιπόν τα τεχνικά ερωτήματα παράλληλα με τους πολιτικούς προβληματισμούς που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Η κυρία Χάουταλα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εννοείται ότι συμφωνώ με όλα όσα είπατε για τις προβληματικές πτυχές του να μην είναι στο ύψος των περιστάσεων ο έλεγχος. Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούω το ότι τώρα στηρίζουμε αυτή τη χώρα που έχει εισόδημα μέσω προς υψηλό. Θα ήθελα να μάθω λίγο παραπάνω πράγματα για τις συνέπειες που αφορούν τις άλλες χώρες του κόσμου. Γιατί μου φαίνεται ότι δεν θα πρέπει να προβαίνουμε σε τέτοιες κινήσεις με τη σημαία της συναντησιακής συνεργασίας. Εκτός αν υπάρχουν κάποιες εξαιρετικές περιστάσεις που είναι τόσο πιεστικές, ε, σοβούν κρίσεις στην χώρα. Τέλος πάντων, τα, διαβάζουμε στις εφημερίδες, αλλά ε, προσοχή να μην ε, καθιερώσουμε έτσι ένα προηγούμενο ατυχές είναι και το θέμα των ναρκωτικών, το θέμα επίσης της ε, ποινής, ε, όλα αυτά ε, επίσης πιέζουν πάρα πολύ. Στη χώρα υπάρχουν τομερά προβλήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις φυλακές κυρίως. Και το πρόβλημα με τα ναρκωτικά έχει σχέση και με τους οροθετικούς, τους ασθενείς του AIDS, πάρα πολύ στις φυλακές. Άρα, μήπως υπάρχει περίπτωση κάπως να το δούμε και αυτό. Γιατί τα ποινωτική σύμφερη φορά, τα βασανιστήρια, τις φυλακές. Το κοινοβούλιο έχει τους πολλές επιφυλάξεις. για εκείνον τον υπερασπιστή των ε, δοκιμάτων γυναικών, ε, πρόκειται για κάποιο δικηγόρο. που υπέστη ότι υπέστηκε. Άρα μήπω γίνεται να τα δούμε και αυτά τα θέματα. Κύριε Σαφχάουτζερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω λόγω να καταγγείλω υποκρισία. Όταν η κυβέρνηση Ομπάμα ε, επιβάλλει κάποιες κυρώσεις ε, ε, για διάφορα θέματα, για τα γεωργικά, για συνεργασία με την χώρα εκείνη. Η Κομισιόν πού ήτανε και ξαφνικά, γιατί τώρα έχουμε κυβέρνηση Τραμπ, μια κυβέρνηση δημοκρατικά εκλεγμένη, βλέπουμε ότι θα διαθέσετε 18 εκατομμύρια. με αυτό δεν σας ε, ε ρεζιλεύει. Τι έγινε αυτό το 40% ε, της, ε, των εξαγωγών μας που πάνε εκεί, την, το Airbus, ε, έχουμε συμφωνίες με τους Κινέζους. Πού είναι η ανεξαρτησία της Ευρώπης όταν ζητούμε την υποστήριξη της ε, Γαλλίας. Εσείς τι κάνατε και τώρα ξυπνήσατε κατά την κυβέρνηση Τραμπ. Τι κάνατε για να υπάρξει η υπεράσπιση της αυτονομίας ως προς τις είπα μα για την τεχνολογία εξαρτώμεθα 100% και τώρα δίνετε τα 18 εκατομμύρια. Τι γίνεται με την τεχνολογία και με τα δολάρια. Δεν θα πρέπει να είστε πιο σοβαροί. Ε, δεν είσαστε. Ποτέ δεν είχαμε ανεξάρτητη πολιτική. Ποτέ δεν ασκήσατε τέτοια πολιτική. Ξαφνικά τώρα λοιπόν ξυπνούμε διότι είναι στην κυβέρνηση ο, ο Τραμπ. Τι λογική έχει αυτή η απόφαση. Είχα πάει με την άφετ στο Ιράν και όταν είπα ότι θα πρέπει να καταληφθεί το δολάριο ε, με κοροϊδεύαν οι συνάδελφοι. Μα αν δεν αποστηνθούμε από το δολάριο δεν θα έχουμε ανεξαρτησία. Ας σοβαρευτούμε και να μην έχουμε, κάνουμε αυτά τα παιχνιδάκια των 18 εκατομμυρίων. Τότε μόνο θα μας πάρουν στα σοβαρά. Ε, δεν ισχύει αυτό όμως σήμερα. Μόνο, μόνο κόντρα στον Τραμπ υπάρχει η παρούσα συνένεση. Ε, αυτοί έχουν συμφέροντα εκείνοι και τα επιδιώκουν, αλλά όχι η Ευρώπη. Βλέπουμε επομένω πόσα πάθη εξάπτει αυτή η συζήτηση, λέει ο Πρόεδρο. Κοιτάξτε, οι κύριοι που μα μιλούν είναι υπάλληλοι είναι και κάνουν ό,τι του λένε πολιτικοί. Είτε των κρατών μελών, είτε ή τη ε, Κομισιόν. Σε άλλου θα πρέπει να τα πούμε αυτά για το πώ λαμβάνονται οι αποφάσει. Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Κύριε Μιλάτη να σου ερωτήσει. Θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι σε εμπιστοσύνη που γίνονται αυτέ οι συζητήσει μεταξύ μα. Δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται και το κοινοβούλιο. Αν έχετε ισχυρά επιχειρήματα, θα μας πείσετε εδώ, γιατί αν δεν μας πείσετε εμάς εδώ, πώς θα πείσετε τους πάρα έξω. Αφού επομένω έχετε την πεποίθηση των απόψεών σας, το θάρρος γνώμη σας και μας τα λέτε, εξηγήστε μας. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το Partnership Fund, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο άλλο τέλος πάντων ταμείο, όπως προβλέπει η συνθήκη. Αυτά θέλουμε να μας πείτε. Το DCI αφορά τη φτώχεια. Πάρα πολλά αιτήματα υπάρχουν κάθε μέρα και περισσότερα για λεφτά από τον προπολογισμό, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι μένουν κάποια λεφτά για τους σκοπούς σύστασης του DCI. Και έχει γίνει αυτό στο παρελθόν. Τέλος πάντων, έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις να απαντήσετε και άλλωστε θα είστε κοντά μας και για το επόμενο θέμα. Και εκεί έχουμε ζητήματα δύσκολα. Για πέστε μας λοιπόν, επί του προκειμένου. Ευχαριστούμε που αναγνωρίζετε το ότι πολλά από αυτά τα θέματα ξεφεύγουν από τη δική μου αρμοδιότητα και θέση. Πώς να σας πείσω όλους. Προσπαθώ να εξηγήσω. τι γίνεται από πλευρά τη Επιτροπή. Ήδη τα έχουμε συζητήσει. Έχουμε διεξαγάγει κατά τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση πολύ καλές συζητήσεις ανά περιοχή, ανά περιφέρεια και με τον Επίτροπο επίσης τα είπατε και έτσι ολοκληρώθηκε η διαδρομή. Άρα να μην θεωρούμε ότι δεν το πήγαμε καλά φέτος, γιατί κάτσαμε και κάναμε μια ε, κάναμε κάποιον απολογισμό για είδαμε τι, τι ισχύει. Τώρα, το ζήτημα είναι το εξής. Το Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι έχει προσβληθεί, ας πούμε ότι έχει προσβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι το αγνόησε η Επιτροπή. Όχι, δεν ισχύει αυτό, Λίντα, σε διαβεβαιώνω. Ε, δεν φοβούμεθα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί επί της ουσίας, όπως σας εξήγησα, ε, ε, αν κοιτάξουμε το, το, το ψήφισμά σας, κάναμε ό,τι λέει. Όχι, όχι, δεν είπαμε για την ε, χρησιμοποίηση του DCI. Όχι, όχι, μιλάω για την ουσία, για το πώς θα κάνουμε τη διαφορά. Έτσι κι αλλιώς αυτά θα τα συζητήσουμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ναι, ναι είπαμε πολλά. και λάβουμε εγώ στο πώς έχουν σήμερα τα πράγματα, το DCI συνεχίζει να ισχύει, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάτι αντίθετο. Ή να σας πω κάτι αντίθετο. Γιατί έγινε αυτή η διαφοροποίηση. Μία από τις αρχές για τις οποίες θεσπίστηκε ο κανονισμός για τον DCI και καλύπτει και αυτή τη διαφοροποίηση, δηλαδή το προβλέπονται εξαιρέσεις παρεκκλήσεις επί τη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Όλα αυτά τα θεσπίζει ο κανονισμός και έτσι δικαιολογούνται οι παρεκκλήσεις ή εξαιρέσεις. Ας πούμε, έχουμε το Ιράκ. Και το Ιράκ έχει μέσα προς υψηλά εισοδήματα και όμως λόγω της ανασυγκρότησης της χώρας δικαιολογεί την χρήση του DCI. Και πολλά άλλα παραδείγματα. Και έτσι και στην Αφρική καταφεύγουμε σε αυτές τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Δεν νομίζω ότι η διαφοροποίηση αποκλείεται απριόρι. Αλλά η νομική ρύθμιση λέει ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Με στενή ερμηνεία κανείς τις επικαλείται και είναι και το σωστό. Και ακριβώ για αυτό το πράγμα και συζητούμε τώρα το τι γίνεται όσον αφορά τέτοια χρηματοδότηση. Όχι, δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει στροφή στην πολιτική μας. Πάντοτε ισχύει αυτό και νομίζω ότι είναι λογική αυτή η τακτική. Τώρα, για αυτά που είπατε σε σχέση με την δέσμευση, τις κυρώσεις, θα τα ξανασυζητήσουμε αυτό την επόμενη φορά γιατί τέτοια θέματα τα βρίσκουμε σε πολλές ε, χώρες, παντού στον κόσμο. Καμπότζη, Μιανμάρ, στο Τατζικιστάν και σε άλλες χώρες. Πολλές φορές πρόκειται για χώρες όπου δεν υπάρχει συμβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτε υπάρχει κράτος δικαίου όπου υπάρχουν πάρα πολλέ ανισότητε. Και άλλα τέτοια. Δεν αρκεί να κουράμε το δάχτυλο, θα πρέπει να εμπλακούμε και να βοηθούμε αυτούς που έχουν ανάγκη βοηθείας. Τους λαούς εκείνων των χωρών δηλαδή. Και πρέπει κάποιος να κάνει την επιλογή. Προσπαθούμε παντού να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν μεταρρυθμίσεις. Μα πώς να υπάρξει ανάπτυξη εάν δεν υπάρχει βοήθεια σε τεχνικό επίπεδο με τα αρμόδια υπουργεία. Γι' αυτό και βοηθούμε για μεταρρυθμίσεις στις χώρες εκεί, τις βαθιές μεταρρυθμίσεις. Πολύ σωστά τα είπατε, ναι, που χρειάζεται κανείς να συνομιλεί με τις αρχές κάθε χώρα. Άρα προσπαθούμε επίσης να επιθετούμε και το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών για να ενθαρρύνουμε και την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει περισσότερο, να μπλέξει περισσότερο η κοινωνία των πολιτών. Μιλήσατε για την μεσονομική στήριξη. Ε, βέβαια, τώρα για το Ιράν δεν συντρέχει κάτι τέτοιο. αλλά έχουμε τα συμπληρωματικά μέτρα, έχουμε τρόπο να μετρούμε τι γίνεται από πλευράς υπηρεσιών του κράτους στις πιο μικρές κοινότητες. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό για τις χώρες εκείνες. Και έτσι σιγά σιγά υπάρχει και υποχρέωση λογοδοσίας από πλευράς διοίκησης κυβέρνησης. Νομίζω ότι έτσι κάλυψα το θέμα του Ιράν ως χώρα ψηλών μεσίων υψηλών εισοδημάτων. Τώρα όσον αφορά το AIDS στις φυλακές, μάλιστα. Ε, ακριβώς όπως και με την ασθένεια εκτό φυλακών σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος είναι κανείς να συνοηθεί, να συνεργαστεί με τις αρχές. Και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες διαλόγου τώρα με την ε, χώρα, με το Ιράν. Έχω ένα μακρύ κατάλογο δεσμεύσεων που υπάρχουν τώρα. Περισσότερες ε, άτυπες, αλλά όμως οδηγούν σε κάποιο υπόμνημα μνημόνιο τεχνικής ε, αρρωγής. Και επίσης υπάρχει συνεργασία για θέματα περιβάλλοντος. Οπότε όσον αφορά και το θέμα του AIDS στις φυλακές, όχι δεν θέλουμε να υπάρχει θεσμενής διάκριση βάρος των εγκλήστων στις φυλακές. Πάντως, είπαμε ότι δεν θα ασχοληθούμε με τα θέματα ασφαλείας, ούτε με το θέμα του εμπορίου ναρκωτικών. αυτά δεν ξέρω τι εννοούσε ο κύριος Σουαφχάουζε στην ερώτησή του απλώς θα σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίζεται βαθύτατα με το τι κάνουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείε. Έχω ασχοληθεί με το εμπόριο, γι' αυτό στα λέω αυτά, αν και τώρα δεν είναι αρμοδιότητά μου. Όλοι με το πρόβλημα είναι τα χρηματοοικονομικά κυκλώματα, οι χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ Ιράν και των υπολείπων χωρών. Τι γίνεται με την εξωτερική πλευρά των κυρώσεων των ΙΠΑ και ξέρουμε τις εταιρείε όπως η Total και άλλες που θέλουν να προβούν σε τεράστιες επενδύσεις. Α, ποια είναι η οικονομική επιτυχία. Και οι επενδύσεις είναι στοχευμένες και επικρίνονται όχι επειδή στο Ιράν, αλλά θα υπήρχαν επικρίσει όπου και να υπήρχε παρόμοια συμπεριφορά. Εμεί χρησιμοποιούμε ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μα. Ε, Ακριβώ επικρίνουμε τον, τον μη σεβασμό των ε, κυρώσεων, του τι κάνουν μέσα ε, Ευρώπης. Ε, βέβαια, οι πολυεθνικέ έχουν συμφέροντα παντού σε όλο τον κόσμο. Τι να ανοιχνεύσει κανείς. Σα σας είπα όμω, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις παρουσίε αρμοδιότητες μου. Θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό οι συνάδελφοι του εμπορίου και των επενδύσεων και φυσικά τα υψηλότερα επίπεδα της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε ξανά με τον Επίτροπο για την ε, διαδικασία ελέγχου. Όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, όπως είπατε, διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή ένα νέο πρόγραμμα για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, στο οποίο ζητείται περισσότερη ευελιξία Γνωρίζω πως είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν αποφάσεις πολιτικού χαρακτήρα που πρέπει να ληφθούν όμως και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δημόσιων πόρων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θα μείνουμε όμως εδώ για να αφήσουμε χρόνο για το επόμενο θέμα το οποίο επίσης είναι αρκετά δύσκολο. Το είπατε και εσείς. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 14, συνεργασία για την ανάπτυξη στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένη της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Μιανμάρ, Φιλιππίνες και Λάος. Μετά το στρατηγικό διάλογο τον Μάρτιο με τον ε, Επίτροπο Μίμητσα, η Επιτροπή μας εξέφρασε αρκετές ανησυχίες για θέματα ε, που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Φιλιππίνες, στο Μιανμάρ, την Καμπότζη και το Λάος. παρέμειναν πολλά ερωτηματικά για την ε, κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες και για τη στάση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής απέναντι σε αυτές. Χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση για να αποφασιστεί η συνέχιση όχι της ε, αναπτυξιακής βοήθειας προς αυτές τις χώρες. Και αυτήν την εβδομάδα είδαμε στις ειδήσει ε, τις έφρικτες παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων των ε, Ροχίνγκια. Γι' αυτό θα ζητήσω από εσά, αγαπητέ συνάδελφοι, να μας ε, δώσετε μία συνοπτική εικόνα της κατάστασης. Εκθέσεις όπως αυτή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αρκετά ενδεικτικές της κατάστασης, αλλά σας δίνω μέσω στο λόγο. Σας ευχαριστώ. Δεν ήξερα σήμερα ότι θα ε, με καλούσατε και σε αυτό εδώ το θέμα, οπότε άφησα τις σημειώσεις μου πίσω. Αλλά φυσικά γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Δεν έχω σημειώσει έτσι κι αλλιώς ε, που να χρειάζομαι. Ναι, ναι, και εγώ ξέχασα τις σημειώσεις μου το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Θεωρώ πως είναι κατάλληλο να ξεκινήσουμε από τη Μιανμάρ. Διότι εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η κατάσταση είναι τραγική. Η διερευνητική αποστολή λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών συναντήθηκε μαζί μου το πρωί σήμερα στις 8.30 και ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα συνάντηση, διότι ακούσαμε μεγάλη προσοχή αυτά που είχαν να μας πούν και νομίζω ότι έγινε συζήτηση ουσιαστική. Και με μεγάλη μου χαρά παρατήρησα ότι υπάρχει κατανόηση της ε, δυναμικής που έχει η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. και τα αποτελέσματα της, ε, και τα πορίσματα της ε, διερευνητικής αποστολής μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ε, συζητήθηκε το θέμα του στρατού στη Μιανμάρ. Η αποστολή είναι πεπισμένη ότι η εξουσία δεν είναι ίσα κατανεμημένη και πως όλα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του στρατού και στην ουσία ο στρατός κάνει αυτό που θέλει όποτε το θέλει. Και είναι πολύ δύσκολο λοιπόν οι πολίτες να ασκήσουν οποιονδήποτε έλεγχο. Και νομίζω αρκεί μόνο να αναφέρω μία λέξη και αυτή είναι η γενοκτονία. Είναι το πιο αποτρόπο έγκλημα που έχουμε εντοπίσει είναι κάτι που διαπιστώσαμε με μεγάλη λύπη. Δεν καταφέραμε καν να πάμε επί τόπου, να πάμε εκεί και τα αποτελέσματα της διερευνητικής αποστολής βασίζονται σε συνεντεύξεις με διάφορους ανθρώπους. Εντοπίσαμε λοιπόν τρία εγκλήματα, το πιο σοβαρό η γενοκτονία. και διαπιστώσαμε επίσης ότι την ευθύνη έχει κυρίως ο στρατός και, άλλες, ε, και άλλοι πέντε φορείς. Τα αποτελέσματα λοιπόν θα παρουσιαστούν στο Συμβουλίο των Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε. Και όπως είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Γκέρενς νωρίτερα, οφείλουμε να συνεχίσουμε ε, τις συνομιλίες με την κυβέρνηση αυτή και να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε ε, στους τομείς ε, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης της υπαίθρου, του επισητισμού, αλλά και σε άλλους τομείς πιο δύσκολους. Ρώτησε για παράδειγμα τι στάση έχουν για τη δράση μας ε, που αφορά τους πολίτες. Ε, μιλήσαμε για τις πρακτικές της αστυνομίας στη Μιαμάρ που χρησιμοποιούν ε, διάφορους τρόπους μη θεμητούς για την αντιμετώπιση των πολιτών. Προσπαθούμε λοιπόν να συζητήσουμε είναι σίγουρα καρυψοκίνδυνο αυτό. διότι τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μιανμάρ. Όμως ακούσαμε ότι είναι θετικά προσκύμενοι στην ε, δράση μας και αυτό που μας είπαν ως ε, συμβουλή είναι ότι θα έπρεπε να δούμε το ρόλο που διαδραματίζει ο στρατός στην οικονομική ζωή της χώρας και να ε, διασφαλιστεί ότι οι οποιασδήποτε κυρώσεις θα επιβληθούν εκεί που πρέπει. Διότι ο στρατός στη Μιανμάρ δεν είναι ένας απλός στρατός, είναι ε, μία γιγάντια οικονομική οντότητα που προστατεύει τα μέλη του και θεωρείται λοιπόν ότι αν επιτεθούμε στο στρατό ε, θα επιτεθούμε και ε, στα συστατικά στοιχεία του. Τώρα νομίζω πως ε, δεν φτάνει ο χρόνος για να μπούμε σε λεπτομέρειες, όμως να πω ότι πέρα από αυτά που είπα, υπερασπίζουμε την ειρηνευτική διαδικασία με τις διάφορες μειονοτικές ομάδες, και φροντίζουμε ε, να διασφαλιστεί μια εξομάλυνση των ε, σχέσεων. Στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις την ειρηνευτική διαδικασία σε πολιτικό επίπεδο. Προσπαθούμε όμως επίσης να ε, παρέχουμε βοήθεια σε διάφορες μειονοτικές ομάδες. Υπάρχει ανάληψη δράση στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα στη Μιανμάρ. Προσπαθούμε να ε, προάγουμε την ισότητα και την ίση πρόσβαση. Είναι πολύ σημαντικό παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση από όλες τις περιοχές και από την Ήπεθρο. Ε, να σας πω επίσης ότι εγώ ίδιο ήμουν στη Μιανμάρ πρόσφατα και παρατήρησα ότι και ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης ελέγχεται από τον στρατό. Υπάρχει ένα Υπουργείο Συνοριακών Υποθέσεων επίσης. Εξετάζουμε με μεγάλη προσοχή το τι συμβαίνει. Εκεί τι συμβαίνει στην εκπαίδευση. Ο στρατός ελέγχει αρκετά ε, ιδρύματα νότα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μιανμάρ. Η απάντηση από την πλευρά της ε, Μιανμάρ ήταν σαφέστατη νομίζω μου. Είπε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η χώρα της χρειάζεται υπουργό συνοριακών υποθέσεων. Υπάρχει λοιπόν δυσαρέσκεια θα λέγαμε μεγάλη για την ανάμεξη του στρατού στις υποθέσεις της χώρας. Ταυτόχρονα όμως, πέρα από όλα αυτά προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που έχουμε στο πλαίσιο συναντήσεων στα Ηνωμένα Έθνη για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας ε, και για να τονίσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας. Και προσπαθούμε να στηρίξουμε τους υπουργούς εκείνους που καταβάλουν προσπάθειες για βελτίωση κατάστασης ε, στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, έτσι ώστε να μην πάνε χαμένες ε, γενιές και γενιές πολιτών ε, που φτωχοποίησαν τη Μιανμάρ, μια χώρα η οποία μετά το τέλος του πολέμου ήταν από τις πιο εύπορες της περιοχής. Και τέλος, μην ξεχνάμε ότι όπως και παντού σε όλη την ε, Νοτιοανατολική Ασία η Κίνα έχει εντονότατη παρουσία και έχει σχέσεις με ε, όλες τις υπηρεσίες της χώρας, όλους τους φορείς και με το στρατό. Και μάλιστα υπάρχουν Κινέζοι πολίτες ε, στη χώρα αρκετοί. Να μην το ξεχνάμε αυτό, διότι φυσικά έχει άμεση σχέση με την ε, πίεση. Αυτά προς το παρόν για τη Μιανμάρ και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις αν έχετε. Ο Σάρλ παρακαλώ ερωτήσεις για τη Μιανμάρ. Θα ήθελα να θέσω και ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με, την, με τις αρχές μας. Ένα θέμα επί της αρχής. Ε, δεν είναι ότι ψηρίζω τη μαϊμού, αλλά θέλω να πω το εξής. Στο πλαίσιο των συμφωνιών μας με τις χώρες ΑΚΕ, αν κάποια στιγμή οι χώρε αυτέ σταματήσουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν στον για παράδειγμα, γίνει πραξικόπημα και έχουν γίνει αυτά. Ε, έρουμε, αναστέλουμε τη συμφωνία συνεργασίας, διατηρούμε την ανθρωπιστική επίγουσα βοήθεια και αποφασίσαμε να αναστείλουμε τις τρέχουσες συμφωνίες και να μην τις εφαρμόζουμε κτλ. Ε, αν λοιπόν η Μιανμάρ ήταν μέλος των χωρών και δεν θα μπορούσατε να κάνετε αυτό που κάνετε τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 95, γιατί αν αναστείλουμε τη συνεργασία για λόγους πραξικοπήματος και δεν τις αναστείλουμε τις συνεργασίες αυτές για λόγους γενοκτονίας, γενοκτονία που αναγνωρίζεται από αρμόδια αρχή, από τον Οργανισμό Εθνών, ε, τότε έχουμε πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Ε, λοιπόν, μεγάλη ιστορία αυτή. Ναι. Ναι, δεν είναι το άρθρο 95, είναι το άρθρο 96 που επιτρέπει, ναι, προβλέπεται μια τέτοια διαδικασία και προβλέπεται στη Συμφωνία Κοτονού ότι μπορεί να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, αλλά είναι διαδικασία, δεν είναι ε, ε, αυτός σκοπός ψοφάκτο. Χρειαζόμαστε γνώμη, γνωμοδότηση από τα κράτη-μέλη. Δεν τη λαμβάνει την αποφασία αυτή η εκτελεστική εξουσία μόνο. Τώρα το να αναστείλουμε ένα ολόκληρο σύστημα, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση. Όχι γιατί θα ντροπιάσει μια κυβέρνηση ή θα δώσει όπλα ε, ε, στα άμεσα οικονομικά συμφέροντα των ελίτ που έχουν πάρει την εξουσία, αλλά γιατί θα βλάψει τους λαούς. Και αυτό το έχουμε δει στην Αφρική πολλές φορές. Το κάνουμε και με πολυθεμητούς και λογικούς ε, λόγους όμως το να αναστρέψουμε αυτή την απόφαση είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Η εμπειρία μας, η εμπειρία μας μας διδάσκει ότι όταν επιστρέφουμε και λέμε ε, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε και να πάψουμε την αναστολή και να ξαναξεκινήσουμε τη συνεργασία, τότε αντιμετωπίσαμε τρομακτικές δυσκολίες. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερον, η ανάπτυξη είναι μια μακροπρόθεσμη ιστορία δεν μπορεί να γίνεται ε, με διακοπτόμενο ρυθμό. Δηλαδή η ιδέα ότι τα αναπτυξιακά κονδύλια, όσα κι αν είναι αυτά, και παρόλο που είναι ανάλογα του προϋπολογισμού του κράτους ε, και παρόλο που μπορεί να λειτουργήσουν ως μοχλός και ως ε, εργαλείο εξαναγκασμού τελικά, αυτό δεν συμβαίνει συχνά γιατί το πιο ισχυρό εργαλείο για ανάπτυξη είναι φυσικά το εμπόριο και έτσι θα ε, αναπτυχθεί η ευρύτερη οικονομία. Τότε στην περίπτωση του Μιανμάρ, της Μιανμάρ, Εάν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσουν ότι θα σταματήσουμε τη βοήθεια στη Μιανμάρ, θα συμβεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το πράξει. Δεν χρειάζεται άρθρο ούτως ή άλλως. Είναι μια πολιτική απόφαση που μπορεί να ληφθεί ανα πάσα στιγμή. Θα ήθελα να μιλήσω για τις συνέπειες των κυρώσεων, των οικονομικών κυρώσεων στη Μιανμάρ πριν από πολλά χρόνια. Αντί να έχουμε στοχευμένες κυρώσεις στα άτομα, να τους εμποδίσουμε από το να ταξιδέψουν, να δεσμεύσουμε τα κονδύλια τους και τα οικονομικά τους και αυτό κάνουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί δεν επιβάλλουν ευρείες οικονομικές κυρώσεις στη Μιανμάρ. Ε, θετούν ορισμένα άτομα, περιορίζουν την κινητικότητά τους και δεσμεύουν τα στοιχεία ενεργητικού τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία εντός ΗΠΑ για ορισμένα άτομα από τη Μιανμάρ μόνο. Εμείς αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ευρύτερε κυρώσεις, μία εκ των οποίων θα είναι και ε, το να σταματήσουμε αυτή την προτίμηση του τα πάντα εκτός των όπλων ε, σαν εμπορική δυνατότητα. Αυτό ισχύει και για την Καμπότζη και για την Καμπότζη. Θα ήταν πρωτοφανές πρεμιέρα για μας να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα έχει όμως ένα γενναίο οικονομικό αντίκτυπο και στη χώρα και στο λαό της χώρας αυτής. Από τη στιγμή που η Μιανμάρ έχει λάβει EBA, ε, βοήθεια τύπου EBA, έχει αναπτύξει μια πολύ σημαντική βιομηχανία φαντουργία, απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και κυρίως γυναίκες. Εάν λοιπόν ανασταλούν και καταργηθούν οι μειώσεις των δασμών. Αυτό θα έχει επιπτώσει στην ευρωπαϊκή αγορά, ε, στο, τις προβλέψεις για, ελεύθερες ελευ... για ελεύθερα ποσοστώσεων και ελεύθερα δασμών και φόρων και πάρα πολλούς ανέργους. ό, ε, όλοι αυτοί θα μείνουν άνεργοι. Και τελικά τι θα κάνουν, θα διασχίσουν τα σύνορα της Ταϊλάνδης και θα γίνουν δούλοι, ήλωτες να δουλεύουν σε εργοστάσια ύποπτα στη Ταϊλάνδη σε βιοτεχνίες που επεξεργάζονται αλλιευτικά προϊόντα. Έχουμε 300 εκατομμύρια ε, μετανάστες χωρίς χαρτιά αυτή τη στιγμή στη Ταϊλάνδη, η πλειονότητα εκ των οποίων είναι από τη Μιανμάρ. Και πρέπει να γνωρίζουμε τι κάνουμε πραγματικά όταν αποφασίζουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στις χώρες και ποιος θα πληρώσει στο τίμημα. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι οι οικονομικές κυρώσεις θα είναι δυσβάσταχτες για τα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας στην κυβέρνηση της Μιανμάρ. Αντίθετα, ο φτωχός λαός της Μιανμάρ είναι αυτός που θα πληρώσει το τίμημα. Αλλά είναι η προσωπική μου άποψη. Κανένα... Ε, δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Είναι δικιά μου προσωπική άποψη. Ο, ο θέλει ξανά το λόγο. Πριν όμως τον δώσω, Κάρολε, να σας ρωτήσω εσάς, θα μιλήσετε και για άλλες χώρες, για την Καμπότζη και τα λοιπά. Ναι, θα επανέλθω. Ο Σάρλ για το θέμα αυτό, ο Κάρολος. Ναι, ξέρουμε πώς λειτουργεί η Συμφωνία του Κοτονού με το άρθρο που διαπιστώ ή τον, τις σοβαρές παραβιάσεις υπάρχει και το άρθρο 96 που επιβάλλεται σκυρός. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Ε, μάλλον δεν χρειάζεται να μας τα πείτε. Εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζουμε όλο ε, και περισσότερες δυσκολίες για να εξηγήσουμε το βεληνικές των κειμένων που αποτελούν τη βάση των συμφωνιών μας. Δεν μπορώ να εξηγήσω σε κάποιον γιατί αναστέλουμε ε, μία ε, συμφωνία συνεργασίας π.χ. με τον Ήγηρα επειδή έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα και δεν το κάνουμε με μια χώρα ε, με την οποία ε, της οποίας ο στρατός είναι αναγνωρισμένα από αρμόδιους φορείς υπεύθυνο ε, για τη γενεκτονία. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια για πήγουσα πρέπει να συνεχιστεί και συμφωνώ, η συμφωνία του Κοτονού δεν το αποκλεί αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι έχει κόστος ε, η πολιτική που υιοθετείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνώ, άρα πρέπει να προσαρμόσουμε τα κείμενά μας και αυτό ισχύει και για την αρχή της διαφοροποίησης, να τα αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα κείμενα και μετά μην τα εφαρμόζουμε. Πώς θα εξηγήσουμε ότι στέκουν αφού δεν φαίνονται να στέκουν. Εάν δεν μπορούμε να εξηγούμε γιατί εφαρμόζουμε τη μία πολιτική στον Ήγυρο και να εξηγούμε τα γιατί εφαρμόζουμε την αντίθετη ε, πολιτική στο, στη Μιανμάρα. Ε, δεν έχουμε καμία αξιοπιστία. Η πρόεδρο μακάρι ο κόσμο τη πολιτική να ήταν απαλλαγμένο από τη διγλωσία. Αυτό είναι αλήθεια. Και από το μία έτσι μία αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, να μιλήσουμε για την Καμπότζη και τις Φιλιππίνες τώρα. Ναι. Καμπότζη. Έγιναν εκλογές. Όλοι εστιάσαν προσοχή μας εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, έγιναν με δημοκρατικές συνθήκες. Με τις αντιπολιτεύσεις φυλακίστηκαν και μπορούμε να πούμε ότι πάρα πολύ πρόσφατα αποφυλακίστηκαν όλοι εκτός από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Και κρεμούν σοβαρές, βαριές κατηγορίες εις βάρος του. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι αυτές οι εκλογές δεν παρέχουν εγγύησεις ε, δημοκρατισμού, ότι δεν είναι δυνατόν να πλαισιώνονται από δική μας ενίσχυση. Την αναστήλαμε, την βοήθεια, την προεκλογική. Και αναστήλαμε τις εκταμιεύσεις, την δημιουργική στήριξη Θέλουμε πρώτα πρώτα να αναλυθεί η πολιτική κατάσταση και τι σημαίνει η δική μας βοήθεια σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Και η Σύμβολη Ανάπτυξης προέβησαν σε σχετική ανάλυση, συνεργαστήκαμε με τους εκπροσώπους μας εκεί, υπέβαλαν αυτή η πρέσβηση τη γνώμη τους. Ε, κατέληξαν στο ότι βοηθά το λαό της χώρας στη συνεργασία. Αλλά αναστήλαμε την ενίσχυση και όσον αφορά την αποκέντρωση όμως ακόμη να λύουμε την κατάσταση και δεν έχουμε στείλει την σχετική ενίσχυση. τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ακόμη επιφυλάσσονται. Για το κατά πόσον η αποκέντρωση έχει επιπτώσεις στην πολιτική κατάσταση. Με δεδομένες τις εκλογές και τις ε, συνέπειες των μέτρων αυτών. Και επομένω με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι δεν θα στηρίξουμε την εκλογική διαδικασία πλέον. Τα ξεκινήσει και πάλι η συνεργασία όσον αφορά την ε, ανάπτυξη, την αλληλεία, τη διαχείριση των ε, δημιουργικών της ε, μεταρρυθμιστή διοίκηση, αλλά όχι ακόμα, όσον αφορά την αποκέντρωση. Πώς να το πω. Είναι δύσκολες οι σχέσεις με τη χώρα σε πολιτικό επίπεδο την τις τη σχέση σχέσεις όσον στον τομέα της παιδείας, των οικονομικών, ε, κοινωνικής πολιτικής, ε, πολιτικής μεταρρύθμισης και πρόσφατα έχουν σημειώσει πρόοδο. Και επίσης το μέτωπο της ανάπτυξης είναι θεματικά τα αποτελέσματα. Ανησυχούμε γιατί αυξάνεται η επιρροή της Κίνας στη χώρα. Η δέσμευση των γιών είναι ζήτημα. Πολύτε γη σε ιδιώτες και αυτό σοβαρό. Όλοι γνωρίζουν τη συνεργασία της χώρας με την Κίνα στα πλαίσια του ΑΣΕΑΝ. Είναι κατά κάποιο τρόπο εκπρόσωπος η χώρα αυτή των κινέζικων συμφερόντων σε αυτή την περιοχή. Οπότε για τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα έχω να πω ότι το πρόβλημα μας είναι το τι πρότυπο δημοκρατής διακυβέρνηση ακολουθούν. Όχι, το πρόβλημα δεν είναι κάθε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούσε κανείς να βρει 10, 20, 50 χειρότερες χώρες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι έχει κατάσταση για την Καμπότζη. Πρόεδρος, δύο λόγια της Φιλιππίνας. Παρακαλούμε σύντομα. Είναι μεγάλος πονοκέφαλος και ίσως είναι καλό παράδειγμα για μια χώρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από το ότι στην Καμπότζη. Και 4.000 είναι οι νεκροί ανθρωποκτονιών και εκτελέσεων χωρίς δίκη. Πρόκειται για αυτόν τον πόλεμο κατά των εργατικών του πρόεδρου της χώρας. Φυσικά και επικρίνεται από τα ευρωπαϊκά Δεσμικά όργανα, ιδίως από το κοινοβούλιο. Οπότε και έχει αρχίσει να στοχοποιεί τα ευρωπαϊκά Δεσμικά όργανα. απειλή κόψει τη συνεργασία μαζί μα. και έχουν υπάρξει και γραφικά στιγμιότυπα στη σχέση μας με τον πρόεδρο του Τώρα εστιάζουν την προσοχή μας σε κάποια σημαντικά μέτωπα προβλήματα στις Φιλιππίνες σημαντικά για όλο τον κόσμο. βοήθεια στο Mindanao προσπάθησα να προκαταβληθούν τόσο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η κοινότητα των μουσουλμάνων δεν θα πρέπει να είναι πηγή τρομοκρατών. Ο Καντάφη βοηθούσε σε αυτή την κατεύθυνση. Ας στο ταμπάο και σε άλλα μέρη. Μπορούμε να δούμε ότι πάλι μπορεί αυτή η περίπτωση της τρομοκρατίας να προκύψει πάρα πολύ εύκολα και πάλι. Κατά τα άλλα, η χώρα σύντομα δεν θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Τελευταία φορά νομίζω έχουμε ένα πακέτο ενίσχυσης. Ήδη επειδή υπάρχει αμυλία απορρόφηση τη χρηματοδότηση, έχουμε συρρυκνώσει την ενίσχυση και, εν πάση περιπτώσει, δεν φρενάραμε στην ε, ενίσχυση, αλλά ο Ε, θεωρητικά, επίσημα, ακόμα την έχει μπλοκάρει τη συνεργασία, αλλά υπάρχουν ε, θετικά σημάδια ότι θα συνεχίσουμε. Ε, επίσης, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, έχουμε καλή συνεργασία με τους αρμόδιους και για την υγεία έχουμε καλή συνεργασία. Βοήθεια προς τους ναρκωμανείς, επανένταξη αυτών και τα σχετικά. Δύσκολο προχωρούμε, αλλά τώρα θα πρώτη μία προσφορά μας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις για τις Φιλιππίνες. Ο κύριος ε, Σαφάουζερ. Θα ήθελα να μιλήσω για τις Φιλιππίνες. Να πω καταρχάς ότι δεν έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στη διπλωματία που προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και περιορίζεται μόνο σε αυτό. Η διπλωματία αυτό που κάνει να διαχειρίζεται συμφέροντα. Το βλέπουμε και με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα και θα πρέπει τα συμφέροντα να ε, συνάδουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν τα εμπιστεύομαι γιατί είναι σαν να κάνουμε νέα, νέου είδους απεικιοκρατία. Πρέπει να στηριχθούμε στην εθνική κυριαρχία των κρατών, να τους πλαισιώσουμε, να τους συνοδεύσουμε ή τότε να πάρουμε την ευθύνη αποσταθεροποίησης και δημιουργίας πραξικοπήματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τους πλαισιώσουμε για να κάνουν ό,τι καλύτερα μπορούν. Γνωρίζω πολύ καλά τις Φιλιππίνες. Πηγαίνω στη χώρα αυτή δύο φορές το χρόνο και έχω πάει και σε διαφορετικές περιόδους στα τέλη της, ε, του καθεστώτος Μάρκος για να τους συνοδεύσω σε αυτή τη ε, δημοκρατική μετάβαση, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο και έχω και πολλούς φίλους και τη γνωρίζω πολύ καλά τη χώρα αυτή. Νομίζω ότι είμαστε υπερβολικά αυστηροί με τον πρόεδρο της χώρας αυτής. Σήμερα η ασφάλεια είναι κάπως καλύτερη. Μπορεί κανείς να περπατήσει στη Μανίλα χωρίς πρόβλημα. Πιο εύκολα από ό,τι στο Παρίσι σχεδόν. Άρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Επίσης ε, έχουν γίνει βήματα στον τομέα της πρόσβασης της υγείας, στον τομέα της εκπαίδευσης, δωρεάν ε, φίτηση για τους μαθητές, για τους φοιτητές. Και μπορεί να μην έχετε ριζοσπαστικέ <laughs> λύσει. Αν έχετε ριζοσπαστικέ λύσει να προτείνετε, να τι συζητήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτερο το Μεξικό και η Κολομβία, με του οποίου έχουμε αγαστέ σχέσει συνεργασία. Δηλαδή, όταν συγκρίνουμε, να έχουμε αποχρώσεις έννοιες, να συγκρίνουμε με το Μεξικό, με την Κολομβία, οι Φιλιππίνες. Ήταν μια χώρα σε σύψη. Και μιλήσατε και για το Ιράν. Υπάρχει θανατική ποινή για όσους υφίσταται το ναρκωτικό. οποίο πεθαίνει από υπερβολική δόση, αυτός ε, υποβάλλεται σε θανατική ποινή. Και πρέπει να δούμε και τις ε, θετικέ πτυχέ. Εάν τελικά ο πληθυσμό στηρίζει τόσο πολύ αυτό το καθεστώς, 90% έστω, και αν αμφισβητούμε αυτά τα νούμερα, ε, εμείς έχουμε πρόεδρο με 35% στήριξη. Είναι, αν ο λαό λοιπόν στηρίζει αυτό το καθεστώς αυτή τη χώρα είναι γιατί βλέπει και τα αποτελέσματα στο επίπεδο τη ασφάλεια που έχει επιτύχει αυτό το καθεστώ. Ευχαριστώ. Σάχλε, ο Κάραλο θέλει κάτι να πει. Ναι. Εν συντομία, κυρία Πρόεδρε, δεν συμφωνώ πολύ με τον κύριο Σαφχάουζερ. Εγώ παραμένω υπέρμαχος της διπλωματίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των ατόμων που έχουν σωθεί. Δεν γνωρίζουμε πόσες ε, ε, περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, γιατί όλα αυτά δεν μπαίνουν στις ειδήσει των 8. Ε, δεν εμφανίζονται εκεί. Η Κίνα δεν επιτρέπει καμία κριτική να τις ασκηθεί σε δημόσιο επίπεδο. Όμως, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αποτέλεσμα του διαλόγου ήταν να δεχθεί η Κίνα ένα δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Ένας ε, Κινέζος πολίτης είχε καταδικαστεί σε θάνατο πρωτοβάθμια και χάρη στις ε, προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφερε οι κινέζικες αρχές ε, να δεχθούν να ε, δικαστεί η υπόθεσή τους σε δεύτερο βαθμό. Άρα υπάρχουν κάποια αποτελέσματα που αξίζουν μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό αξίζει να έχουμε διπλωματικά διαβήματα. Ναι, απολύτως, ναι, κύριε Σαφχάουζερ. Είναι επίπονη διαδικασία, είναι χρονοβόρα, είναι κουραστική, είναι αυστηρή, είναι σκληρή, είναι δύσκολη, αλλά είναι απαραίτητη. Η διπλωματική άγουσα. Ξέρετε, παλιά με το, την εποχή του σιδηρού παραπετάσματος μπορούσε κανείς με απόλυτη ασφάλεια να περπατήσει στη Μόσχα. Υπήρχε ασφάλεια τότε, σίγουρα. Ο κύριος ήθελα να ρωτήσω για τα καταπήγοντα, κάτι που χρησιμοποιούμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα καταπήγοντα είναι ένα μέσο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε παρόμοιες περιπτώσεις όπως στη Μιρανμάρ, στις Φιλιππίνες κτλ. Ε, ποια είναι η εμπειρία σας από, ε, αυτό, από τη χρήση του μέσου αυτού. Έχει κάποια χρησιμότητα υπήρξαν και κάποια πολιτικά σχόλια στις ερωτήσεις αυτές, οπότε μπορείτε να επιλέξετε τι θα απαντήσετε. Θεωρώ πως υπάρχει πράγματι διαφορά μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιεί κανείς. Εξαρτάται από το τι θες να χρησιμοποιήσεις. Η πρώτη μου θέση ήταν στο Βιετνάμ και το 1996 ο κατάλογος των πολιτικών ε, κρατουμένων ήταν τεράστιος και έπρεπε να συνομιλήσουμε και με τους ε, Γάλλους, τους Βέλγους, με όσους ήταν εκείνη την εποχή παρόντες στη χώρα. Θεωρώ λοιπόν πως ε, είναι αποτελεσματικό αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την διπλωματία. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τοποθετούνται για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάποια χώρα και ε, αυτή είναι μια πολύ ε, λεπτή ε, πολιτική κίνηση Η αναφορά δηλαδή σε θύματα, σε παραβιάσεις, σε διεθνείς οργανισμούς. Φυσικά υπάρχουν και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά ελέγχονται από τις χώρες εταίρους μας και φυσικά έχουν αντίκτυπο, ασκούν πίεση, όμως έχουν και κάποιο κόστος οι πρέσβεις μας στις χώρες αυτές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις. όλων αυτών των ψηφισμάτων, των αποφάσεων, των δηλώσεων. Στις Φιλιππίνες, λοιπόν, Πιστεύω ότι, για να σας πω και την άποψή μου, υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα και έχω μιλήσει με διάφορους πρέσβες στη Μανίλα, έχω ακούσει για το πόσο επιθυμούν μια εξομάλυνση της κατάστασης, ε, αν έχει κάποια αξία αυτό, ακριβώς ε, γιατί υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις στη χώρα από την Ευρώπη. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, διότι υπάρχει κίνδυνο σταδιακά επενδύσεις αυτές να αντικατασταθούν από κινέζικες επενδύσεις. Μάλιστα, νομίζω πως ε, αρκετά σας ταλαιπωρήσαμε, σας είχαμε μία ώρα και 45 λεπτά και σας εκτοξεύαμε ερωτήσεις μία μετά την άλλη. Νομίζω πως δεν έχει φυσικά τελειώσει το θέμα εδώ. Λαμβάνουμε συνέχεια επιστολές από πολίτες που μας ζητούν εξηγήσει για το τι συμβαίνει. Ε, αυτά που είπε και ο Σάλ Γκόρενς δηλαδή. Νομίζω πως ε, οι απαντήσεις που μας δώσατε ήταν ικανοποιητικέ και σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για αυτά τα δύο σημεία. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, ομάδα για την ε, Μέση Ανατολή που παρότι μας στήριξε αριθμητικά δεν μπόρεσε να ακούσει την ανάλυση μας για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Okay, we go on. Μάλιστα. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο για σήμερα, πριν τους ε, συντονιστές, το σημείο 15, ΠΟΕ, η συνέχεια. Η Επιτροπή Εμπορίου συντάσσει μια έκθεση για το μέλλον του ΠΟΕ. Όπως γνωρίζετε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι ένας διεθνής οργανισμός που ε, επιβλέπει και ελέγχει τους ε, κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση από πολλές ε, κατευθύνσεις και από την αριστερά αν θέλετε αλλά και πρόσφατα από τον ε, πρόεδρο Τραμπ ο οποίος έχει ασκήσει κριτική στον ΠΟΕ όπως και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Φυσικά όλα αυτά έχουν και αντίκτυπο διότι ενώ αποδυναμωθεί ο ΠΟΕ τότε θα έχει αυτό επιπτώσεις και στις πιο αδύναμες χώρες. Δεν θα μπορούν πλέον να ε, έχουν άποψη. Αλλά για αυτά θα δώσω το λόγο στην κυρία Σάντζες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι η Επιτροπή μας να συντάξει ε, γνωμοδότηση για το μέλλον του ΠΟΕ. Το εμπόριο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και οι εμπορικές πολιτικές όποιου χαρακτήρα και αν είναι και όποιες φύσεις και αν είναι επηρεάζουν την ανάπτυξη και την αναπτυξιακή πολιτική. Και η δική μας Επιτροπή και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα, πρέπει να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα αυτό το εγχείρημα και να προσπαθήσουμε να ευθυγραμμιστούμε με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απέτηση να, υπάρχουν συνοχή, να υπάρχει συνοχή στις ε, ε αναπτυξιακές πολιτικές. Η απελευθέρωση του εμπορίου δεν είναι αποφασιστική για τη μείωση των ε, ανισοτήτων. Αντιθέτως, αν υπάρχει υπερβολική απορρίθμιση, ο αντίκτυπος είναι πολύ αρνητικός στη ζωή των γυναικών ή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε τον ΠΟΕ, ο οποίο είναι ένα φόρουμ πολυμερούς διαπραγμάτευσης και είναι χώρος όπου μπορούν να μπουν κανόνες στο διεθνές εμπόριο και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει τον εκδημοκρατισμό του Παγκόσμια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου για να γίνει πιο νομιμοποιημένος οργανισμός και να ακουστούν όλες οι φωνές σε αυτό το φόρουμ. Θα πρέπει να έχουμε εμπορική πολιτική ατζέντα με βάση ένα πιο δίκαιο εμπόριο προς όφελος όλων. Η ανάπτυξη τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας και να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών χαμηλού εισοδήματος. ΠΟΕ οφείλει να αναγνωρίσει ξεκάθαρα το ρόλο που μπορεί να διαμαδραματίσει το εμπόριο για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει ο ΠΟΕ γι' αυτό το λόγο να αξιοποιήσει ω ελάχιστο πλαίσιο, ω ελάχιστη βάση εργασία τη Συμφωνία των Παρισίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες δεν πρέπει να δίνουν λάβη για κατακαιρματισμό. Δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τα δημοκρατικά ε, φόρουμ όπου ε, αυτά είναι αυτά που θα πρέπει να ρυθμίζουν το παγκόσμιο εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να θεμελιώσουν τον εκδημοκρατισμό ε, του παγκοσμίου εμπορίου. Τα μέλη του ΠΟΕ θα πρέπει να εγγυηθούν τη δημοκρατική νομιμότητα και τη διαφάνεια την κοινοβουλευτική διάσταση αυτών των οργανισμών και αυτές είναι, αυτά είναι τα βασικά αιτήματα που θα παρουσιάσουμε στο προσχέδιο γνωμοδότησής μας και ελπίζουμε με να τύχουν επιτυχία στην Επιτροπή σας και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν σύντομοι και σαφείς. Ο κύριος και ο κύριος Νόιζε και μετά ο κύριος Αφχάουσερ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα την συγγήτρια για την γνωμοδότηση. Θεωρώ πως η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ θα διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην άσκηση πολιτικής στο μέλλον γνωρίζουμε ότι αυτή η συζήτηση λαμβάνει χώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλιστα τα αρχικά αποτελέσματα των διαβουλεύσεων ακριβώς εξαιτία των ΗΠΑ δεν οδήγησαν πουθενά. Θεωρώ ότι η δημιουργία της ε, κοινοβουλευτικής ε, συνέλευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ε, με τον Πατρίκ Ήμασταν υπεύθυνοι για την επίβλεψη του όλου εγχειρήματο και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει μεταξελιχθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, οι ευρωβουλευτές να συμμετέχουν στην ε, συζήτηση για το μέλλον του ΠΟΕ. αλλά είναι και πολύ σημαντικό η αντιπολίτευση να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Πολλές φορές ε, οι κυβερνήσεις έχουν ε, ιδιαιτερότητες στην ισορροπία των ε, δυνάμεων. Πολλές φορές ένα κυβερνητικό σύστημα είναι όμως πονδιακό, οπότε και εκεί υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπάρχει λοιπόν διαφορά στο, στα επίπεδα συμμετοχής. Υπάρχουν ε, λοιπόν κάποια σημεία στα οποία θα ε, πρέπει πιστεύω, πιστεύω να σταθούμε. Στην διευκόλυνση του εμπορίου, για παράδειγμα, είναι κάτι πρέπει να στηρίξουμε και ε, οικονομικά και με ανθρώπινο δυναμικό. Ε, διασυνοριακό εμπόριο επίσης είναι ένας τομέας που πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό να προσέξουμε, διότι και εκεί υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα. Μετά, ε, εμπορικές διαφωνίες. Είναι ένα τομέα ο οποίο πέρα από τη διευκόλυνση του εμπορίου μπορεί να διαταρματίσει εξίσου σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό οφείλουμε να αναμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το Aid for Trade να φροντίσει για την ε, περαιτέρω ανάπτυξή του θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο ε, το οποίο θα δίνει προσοχή και στήριξη στην βιώσιμη ανάπτυξη, στη, στα ασφαλή τρόφιμα, ε, ασφαλή ε, ίδρυυση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτές είναι οι κεντρικότερες και σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φτωχότεροι. Γι' αυτό νομίζω πως δεν πρέπει να ξεχνάμε και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε. Επίσης, δεύτερος πυλώνας, ε, ε, τρίτος πυλώνας, μας συγχωρείτε, ε, γεωργία. Είναι πάρα πολύ σημαντική για τον επισητισμό. Χρειάζεται, να υπάρχουν οικονομικά ασφαλή τρόφιμα προσβάσιμα. Ε, μάλιστα πρόσφατα είδα και μια καρικατούρα που νομίζω είναι ενδεικτική, μια Αφρικάνα η οποία κρατά στο χέρι της μία ε, ντομάτα που της κόστησε ένα ευρώ και δίπλα της ε, μία Ευρωπαία νοικοκυρά με ένα καλάθι ντομάτες που κόστησε το ίδιο. Αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην ε, Αφρική για παράδειγμα και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και νομίζω πως πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας έτσι ώστε να διορθωθεί. Πρέπει να γίνει πιο ελκυστική η πολυμερής προσέγγιση. Ήδη στο Buenos Aires κατέστησα φες ότι χρειάζονται ε, ριζικές μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια ε, για το ότι έβαλε στο προσκήνιο το θέμα της αναπτυξιακής πολιτικής. Νομίζω πως η γνωμοδότηση πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νόιζερ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για τη γνωμοδότηση εκ μέρους, ε, του, Φράντσο, του κυρίου Φρουντζουλίτσα, ο οποίος δυστυχώς ε, απουσιάζει σήμερα. Η γνωμοδότηση λοιπόν πολύ σωστά δίνει έμφαση στη λειτουργία, στην εύρυθμη λειτουργία του ΠΟΕ ως ένα ε, φόρουμ διαπραγματεύσεων και ανοιχτή συζήτηση για θέματα που αφορούν το εμπόριο. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε την θετική συνεισφορά του Fair Trade στην ε, ευημερία. Χρειάζεται λοιπόν να ζητήσουμε ένα σύστημα ίσο για όλους. 32 κράτη-μέλη του ΠΟΕ αυτή τη στιγμή είναι αναπτυσσόμενες χώρες και πρέπει ε, να δώσουμε τη δυνατότητα στις χώρες αυτές να έχουν πρόσβαση σε ανοιχτό εμπόριο και να ανταμείβονται οι ε, προσπάθειές τους. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα μέλη του ΠΟΕ που ε, είναι αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν να ακολουθήσουν βήματα απελευθέρωσης του εμπορίου χωρίς να είναι υποχρεωμένα να ε, αναλάβουν περισσότερα από αυτά που μπορούν. Πρέπει οι, δεσμεύ, οι υποχρεώσεις να είναι ανάλογες της ε, δυνατότητας του κάθε κράτους. Επίσης, οι συμφωνίες διευκόλυνσης του εμπορίου είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες απολαμβάνουν ε, μέτρα προσαρμοσμένα στις δικές τους ε, δυνατότητες έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν τη συμφωνία. Ο ΠΟΕ μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν την μείωση της φτώχειας, την υγεία, την παιδεία με τη στήριξη εμπορικών μεταρρυθμίσεων υπέρ της ανάπτυξης και υπέρ του εμπορίου. Επιπλέον, το πολυμερές πλαίσιο του ΠΟΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των αναγκαίων ευέλικτων μέσων για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Τέλος, προς αύξηση της ε, διαφάνειας και ε, για να εγγυηθούμε την ε, ομαλή συνέχεια του διεθνούς εμπορίου πρέπει να ε, επιμείνουμε στην ε, έντονη κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μεταρρύθμισης του ΠΟΕ για να καταστεί πιο αποτελεσματικός με μεγαλύτερη διαφάνεια και τέλος θα ήθελα και ο συνάδελφος Φουντζουλίτσα να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκόρντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και συμφωνώ με τα περισσότερα που αναφέρονται στην γνωμοδότηση. Να σκεφτούμε μήπως ε, κάνουμε έτσι ένα δωράκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ο πρόεδρος της ήρθε σε επαφή με τον πρόεδρο τον είπα χωρίς να έχει φήμη φανατικού της ακρόασης και τι έγινε τότε μπόρεσε να μιλήσει εκ μέρους των 27 έτσι γι' αυτό τα κατάφερε να μιλήσει με τον μεγαλύτερο εκπρόσωπο της Αμερικανικής πολιτικής. Τίποτα ακόμα δεν έχει κλείσει, τίποτα δεν είναι βέβαιο, αλλά αυτό που έγινε είναι σημαντικό. Αυτά σας τα λέω, γιατί υπάρχουν πολλά ενισχυτικά που συμβάνουν. Είπαμε για την προηγούμενη παρέμβαση, για το όργανο επίλυσης διαφόρων. Εκεί έχει επτά δικαστές. Τώρα τέσσερις υπάρχουν, των τριών η θητεία δεν ανανεώθηκε. Αν είναι κατά της ανέωσης θητείας η Αμερική, για τον τέσσερο ας πούμε, τον τέταρτο ας πούμε, αν γίνει κάτι τέτοιο, μα τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το όργανο επίλυσης διαφόρων. Μα αυτό είναι από τα βασικότερες κατακτήσεις του πολυμέρους οργανού, να, έχει καθαρά δικαστικό χαρακτήρα. Οπότε καλά τα πάει η Κομισιόν. Μπράβο της. Δεν ναι, είναι θέμα διμερών συμφωνιών. Είναι για το ότι όλοι αυτοί επιτέθηκαν στο πολυμερές εμπόριο. Α, είδατε τι έγινε με την ε, πνευματική ιδιοκτησία, τα φάρμακα για τις αντισώμενες χώρες, εντάξει, αυτά καλά πήγανε, τα υπόλοιπα όμως μπλοκαρίστηκαν. Ε, τώρα πάμε για διμερεί συμφωνίες. Εάν το εν λόγω όργανο επίλυσης διαφορών δεν μπορεί πλέον να συνεδριάσει και να κρίνει. Άρα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. τι θα γίνουν οι συμφωνίες που συνάπτονται α, ε, στα πλαίσια του ΠΟΕ. Έχουμε και τις καταγγελίες των αδειωμένων χωρών. Περίπλοκα τα πράγματα. Αλλά μπορεί να υπάρχει μια ακτίνα ελπίδας. Η Ευρώπη μπορεί να σώσει την κατάσταση. Ευχαριστούμε. Σαφχάζ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, όποτε είναι σαν τον ΟΗΕ, διεθνής οργανισμός. Στην αρχή ήταν λόμπι για το διεθνές εμπόριο και υποστηρίζεται από είπα γιατί της ε, συμφέρει. Γιατί ήθελαν τον ε, πόλεμο να κυριαρχήσουν οικονομικά. Και ο οργανισμός τούτος όταν σταμάτησε να εξυπηρετεί όταν κατέληξε να είναι ο πρώτος εταίρος η Κίνα και ούτω η ΙΕ να βοηθήσει τις απώλειες του βιομηχανικού μέτωπο, ε, τότε αποφάσισαν είπα να δυναμητήσουν τον ΠΟΕ. Και εγώ συμφωνώ με αυτό. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει εδώ και καιρό. αντίθετα με τον ΟΗΕ είναι λόμπι, δεν είναι διεθνής οργανισμός ο ΠΟΕ. Δεύτερον, ενίον νόμισμα και ε, η αγορά κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Είδατε τι γίνεται με τους Γερμανούς και την Ευρωζώνη. Όλοι που είναι στην Ευρωζώνη τα πάνε χειρότερα. εκτό από αυτού που είναι εκτό Ευρωζώνη, και έχουν ελεύθερη διακύμανση. Αν είδατε τι γίνεται με Πολωνία, Ουγγαρία, την Ανατολική Ευρώπη. Βλέπετε επομένω το ότι η αγορά ευνοεί του ισχυρού και αδυνατίζει τους πλέον αδυνάμου. Αυτό είναι η τρίτη παρατήρηση. Το 48 την απάντησαν τον εγώρος και είπαν ότι τα πλεονάσματα όπως και τα ελλείμματα δεν είναι κάτι καλό για το βιώσιμο εμπόριο. Χρειάζεται ένα δίκαιο εμπόριο. Δεν θα πρέπει το εμπόριο να οδηγεί ε, στο να κάνει κάποια χώρα πιο φτωχή και να τη πλήσει την ε, κυριαρχία. Αυτό που λέμε μερκαντιλιστικό πρότυπο. 280 δις είναι το εμπορικό πλεονάσμα της Γερμανίας. 450 της ε, Κίνας. Είδατε, πέρασαν την Κίνα όσον αφορά την κατακεφαλή αναλογία. Μα γι' αυτό και στέφτηκα τη Γερμανία ο Τραμπ. Και έχει δίκιο. Νομίζω ότι το οικονομικό μοντέλο που ακολουθούμε είναι αυτοκτονικό. Εάν θέλουμε αυτό να έχουμε ως βάση για την οικοδόμηση της Ευρώπης, ε, τότε η Ευρώπη θα εκραγεί. Ούτε υπάρχει κανένας μηχανισμός ελεγγύης, γιατί θέλουμε την αγορά, αλλά δεν θέλουμε μηχανισμό αλληλεγγύης. Να έχουμε ευρώ και να έχουμε κάτι που να ε, αντισταθμίζει. Αλλιώς να μην το έχουμε το ευρώ και έτσι θα χαθούν αυτά τα 800 δίστα γερμανικά. Έτσι είναι τα οικονομικά. Εσείς κύριε Ρουμπίχη. Τι θέλετε να πείτε. Όχι, όχι. Δεν είναι, δεν είναι Γερμανός. Α, ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, αλλά εδώ και πολύ καιρό τα λέμε αυτά για όλες τις ευρωπαϊκές ε, οργανώσεις και οργανισμούς. Δεν είναι θέμα γαλλικό να κάτσουμε και να προβληματιστούμε σε σχέση με το οικονομικό μας πρότυπο και μοντέλο. Ακολουθούμε τον φιλελευθερισμό, όμως δεν ξεκίνησε έτσι η Ευρώπη. Πάντοτε έχει προτεραιότητα η συνεργασία, όχι ο ανταγωνισμός, αλλά εμείς κάναμε τον ανταγωνισμό Θεό και εκπλησόμεθα γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ούτε αλληλεγγύη υπάρχει επίσης now Και τώρα ο κύριος Μαρσελέση, ο οποίος παρά το όνομά του δεν είναι Ιταλός. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε και την ε, Λόλα που σύμφωνα με την κατεύθυνση της γνωμοδότησης. Οπότε έτσι θα πρέπει να εμβαθύνουμε, συμφωνούμε, υπενθυμίζουμε ότι η απελευθέρωση της αγοράς δεν είναι κάτι που αποτελεί αυτό σκοπό ή κάτι που είναι θετικό από μόνο του. Θα πρέπει να δούμε αν κάνει κάτι για την ενημέρωση της φτώχειας και το περιβάλλον και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθηθεί το πολυμερές επίπεδο συναλλαγών. Έχουμε τώρα τον τελευταίο γύρο αυτών των συμφωνιών που θέλουμε να μην είναι διμερείς και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να εκδημοκρατιστεί ο ΠΟΕ. Τώρα δεν διακρίνεται από μεγάλη διαφάνεια. Πρέπει να εκδημοκρατιστεί περισσότερο. Επίσης, κυράρχηση των κανόνων. Συμφωνούμε. Το πιο σημαντικό δεν είναι το εμπόριο, δεν είναι το εμπόριο αυτός σκοπός. Το θέμα είναι υπάρχει ευημερία για τον κόσμο μέσω του εμπόριου σε όλο τον πλανήτη. Άρα αυτό είναι κάτι όπως το θεματολόγιο του 2030 που σημαίνει τον Παρισιών που είναι πάνω από το εμπόριο. Δεν θέλουμε εμπορικέ συμφωνίες που να αντιβαίνουν τι ε, συμφωνίες των ε, Παρισίων. Το εμπόριο θα πρέπει να βοηθά περισσότερη βιωσιμότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Άρα θα πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο αυτά τα οποία μας επισήμανε η συγγήτρια και θα δούμε τι γίνεται με τη δυσμενής διάκριση για τις μεθόδους παραγωγής, για κάποια προϊόντα, κάτι το οποίο συμβαίνει στον ΠΟΕ. Θα δούμε τι γίνεται με το αποτύπωμα του άνθρακα, να δούμε πώς αυτό θα βοηθήσει να είναι τα πράγματα πιο δίκαια και αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα από τον ΠΟΕ. Και έτσι υπάρχει μια λυσίδα αξίας και για τα κλώσσα φαντουργικά. Επίσης η αρχή της προφύλαξης είναι βασική αρχή και για το εμπόριο να αναγνωριστεί, να κατοχυρωθεί αυτό. Και μεταφορά τεχνολογίας, που να μην βλάβει το περιβάλλον, τρίψ, ντόχα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος, όλα αυτά να αναδειχθούν μέσα στον πόλεμο. βιοπικιλότητα, βιοπειρατεία που αναδείχθηκε τώρα στον αιώνα μας και να αναγνωριστεί παντού στον πλανήτη το εμπόριο να μην είναι αυτός σκοπός, να είναι μέσο για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή ευημερία για όλους. Λόλα, έχεις τίποτα να προσθέσεις? Α, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτη. Περιμένουν τη σειρά τους υπομονετικά. Λιτκόφσκι. Και ο κύριος Πούζα. Από την Γενική Διεύθυνση Εμπορικών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια γενικά σχόλια και μετά κάποια πιο ειδικά. Με την τελευταία παρέμβαση να ξεκινήσω να επαναλάβω σε όλους τους τόνους ότι είναι πολύ αληθές και σαφές ότι το εμπόριο δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι κάτι που προέρχεται από την συμφωνία του ΠΟΕ. Πρώτος στόχος της σύστασης αυτής του, αυτού του οργανισμού είναι η οικονομική ανάπτυξη των μελών και η επιδίωξη αυτού του στόχου. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η οργάνωση αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει ποτέ αντιμετωπίσει. Σήμερα τις αντιμετωπίζει αυτές. Και αυτοί που θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι τα πιο αδύναμα και τα πιο φτωχά μέλη του ΠΟΕ, οι χώρες αυτές. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία και να ε, αφήσουμε πια αυτή την κρίση. Η Επιτροπή έχει καταλήξει σε ορισμένες ιδέες για τη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Κάποιες από αυτές τις ιδέες τις έχουμε μοιραστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλούμε για το ε, θέμα της παρακολούθησης, της εποπτείας, το θέμα της διευθέτησης, ε, της επίλυσης των κρίσεων και των διαφορών θα έχουμε πλήρη παράλυση πολύ γρήγορα αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα των ε, αρμοδίων φορέων. Χαίρομαι λοιπόν που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Πρώτον. Δεύτερον, ως προς τον αντίκτυπο της απελευθέρωσης του εμπορίου. Στόχος του ΠΟΕ είναι να στηρίξει την ανάπτυξη των μελών του στην ιστορική του διαδρομή αλλά και τον προκάτοχό του που ήταν η ΓΚΑΤ, η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, είχαμε άριθμα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο το εμπόριο είχε θετικό αντίκτυπο και η ανάπτυξη του εμπορίου είχε θετικό αντίκτυπο στην, στις χώρες και ότι ε, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχεια με αυτόν τον τρόπο. Δόθηκε το παράδειγμα της Καμπότζης και των, ε, του προτιμησιακού καθεστώτος που απολαμβάνουν και πώς αυτό τους βοηθάει στην οικονομική τους ανάπτυξη. Ως προς τις πολυμερείς και διμερείς εμπορικές συμφωνίες θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι Όλες αυτές οι συμφωνίες συνάπτονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ο οποίος προβλέπει τέτοιου είδους ε, συμφωνίες, γιατί επιτρέπουν στα μέλη να επιδιώξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να εμβαθύνουν στις προσπάθειές τους. Μπορούν να δημιουργήσουν έτσι οι κανόνες και οδηγούν σε ακόμα περισσότερες πολυμερείς συμφωνίες. Σας θυμίζω τις διαπραγματεύσεις ε, για τα περιβαλλοντικά θέματα. Ήταν πολυμερής ε, διαπραγμάτευση αυτή. Σας θυμίζω και τις διαπραγματεύσεις για την ε, τεχνολογία ε, ε, της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Τώρα, σε σχέση με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι πολύ σημαντικό που ένα συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων. Και αυτό φάνηκε και στο έγγραφο. Μπορεί ο ΠΟΕ να συμβάλλει ιδιαιτέρως, να ενισχύσει τις, ε, εξαγωγές, να ε, εξαλείψει τις ενισχύσεις στην αγροτική πολιτική, ε, οι ενισχύσεις στην αλία. Κάνουμε εκεί διαπραγμάτευση, γίνεται διαπραγμάτευση εντός του ΠΟΕ. Και όλα τα μέλη αναγνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η εντολή που έδωσαν οι ηγέτες το 2015, δηλαδή να συνεχιστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις και να εξαλειφθούν οι πιο επιβλαβείς ενισχύσεις ε, στην αλλιευτική δραστηριότητα. Και από πλευρά ΔΕΦΚΟ, Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ για την Ανεπτυξιακή Συνεργασία, δύο λόγια θα ήθελα να πω. Το Aid for Trade, βοήθεια για την ανάπτυξη, για το εμπόριο, εμείς ε, έχουμε εκδώσει ανακοίνωση για το θέμα αυτό τον περασμένο Νοέμβριο και με ένα μήνα μετά είχαμε τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα Aid for Trade, βοήθεια για το εμπόριο, διότι ε, το εμπόριο δημιουργεί ευκαιρίες σε πολυμερές και διμερές επίπεδο και αντισταθμίζει τις προκλήσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση και την ε, όλο και μεγαλύτερη διεθνοποίηση. Έτσι έχουμε και καλύτερες σχέσεις μεταξύ ε, εμπορίου και ε, επενδύσεων, γιατί έτσι διαφοροποιούνται οι οικονομίες. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουμε σε αυτή τη συζήτηση. Αναφερθήκατε στη διευκόλυνση του εμπορίου και αυτό το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ξέρετε, ε, το 2014 όταν κάναμε τις ε, διαπραγματεύσεις για το TFA, η Επιτροπή δέσμευσε 400 εκατομμύρια ευρώ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, για το Trade Facilitation Agreement, από τη στιγμή που θα τίθετο σε ισχύ η συμφωνία και μετά. Αλλά έχουμε ξεπεράσει αυτές τις δεσμεύσεις. Έχουμε ε, κάνει πολύ μεγαλύτερες πληρωμές. Και αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. για τη διευκόλυνση του εμπορίου και της εμπορικής δραστηριότητας είναι και ο τρόπος να διασφαλίσουμε ότι κάποια μέρη του πληθυσμού που ασκούν εμπορική δραστηριότητα κοντά στα σύνορα θα μπορούν να κάνουν εμπορικές αναλλαγές απρόσκοπτα. Και είναι μια λύση για την Αφρική αυτή να έχουμε συμφωνίες όπως η Τριμερή Συμφωνία ή η Αφρικανική CF να ε, λειτουργήσουν αυτές οι συμφωνίες και να εφαρμοστούν και να είναι αποτελεσματικές. Η Λόλα για τα καταληκτικά σχόλια, παρακαλώ. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ τους κοιόδης εισηγητές, εξ όσων ε, κατάλαβα ε, και εξ όσων άκουσα, θεωρώ ότι κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί θα μπορέσουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Για να δω τις σημειώσεις μου, καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 3 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Με αυτά και με αυτά λοιπόν ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Σας χαιρετώ όλους. Θα έχουμε τώρα συνεδρίαση των συντονιστών που θα ξεκινήσει σε 5 λεπτά. Οι συντονιστές εδώ σε 5 λεπτά, οι υπόλοιποι μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Ευχαριστώ.